Uh, Καλημέρα σας. Η κυρία Ματσόνη θα καθυστερήσει. Θα είναι σύντομα πάντως μαζί μας. Συνεπώς θα αυτοσχεδιάσω λίγο Περνάμε στο σημείο 1, έγκριση του σχεδίου μερίσιας διάταξη. Ο κύριος Γιάρ δεν είναι σήμερα μαζί μας, συμμετέχει σε μια επίσημη αντιπροσωπεία της Επιτροπής Γεωργίας. Επομένως, ζητά συγγνώμη για τη σημερινή του απουσία. Θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες όταν φτάσει στην αίθουσα η κυρία Ματσόνη. Όπως σας είπα, θα φτάσει πολύ σύντομα. Το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης έχει να κάνει με τις ψηφοφορίες για διάφορες εκθέσεις τις οποίες έχουμε συζητήσει και σχετίζεται επίσης και με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Όσον αφορά τις αναφορές για τη σημερινή συζητή... συνάντηση, θα ήθελα να ενημερώσω ότι το σημείο 11 θα παρουσιαστεί από τον κύριο Κρεσέντο και από τον κύριο Μπαρμπαρίνο το σημείο 12 θα παρουσιαστεί από τον κύριο Πέσκοτ και Σίφρεντ για το συγκεκριμένο σημείο ένας ο κύριος Χριστοφόρης από την Κυπριακή Προεδρία, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Προεδρία, θα κάνει μια δήλωση για το σημείο 15 θα παρουσιαστεί από τους Μαρινέλα και Μπερτούτσι. Συγγνώμη κάνω λάθος με το κύριος και το κυρία. Το σημείο 16 από την κυρία Ροκόφκασκα και τον κύριο Μπάρσκι και το σημείο 19 από τον κύριο Γουάν Λόπες de Είναι παρόν επίσης ο αναφέρον για το σημείο 19, το οποίο θα παρουσιαστεί μετά το σημείο 16. Δεν ξέρω πώς, τι άλλο μπορώ να κάνω για να σας κρατήσω ξύπνιους, όχι δεν μπορώ να τραγουδήσω, συγγνώμη. Μου πρότεινε να τραγουδήσω ένα τραγούδι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πάντως με την ψηφοφορία. Πρέπει και εγώ να φύγω βέβαια γιατί πρέπει να πάρω ένα αεροπλάνο σε μία ώρα. Δεν ξέρω, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Είναι πολιτικά ορθό να κάνουμε κάτι τέτοιο. I know, we all know that. I have my own, I understand that. Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πάντως αν μπορούμε τυπικά, επισήμως, να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις προφορίες χωρίς την παρουσία της Προέδρου. Μάλιστα, ωραία. Αν διαδικαστικά δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα... I vote as well. Okay. So we start with uh, the annual report of the activities of the Committee on Petitions. Ξεκινάμε με την ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών για το έτος 2011. Ο κύριος Τσίτσεστερ ενδεχομένω θέλει το λόγο. Όχι, δεν θέλει το λόγο. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσίτσεστερ που δεν παίρνετε το λόγο. Ξεκινάμε με τη συμβαστική τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αποχές, συγγνώμη. Δεν υπάρχει καμία αποχή. Με συγχωρείτε, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ψηφοφορίες προεδρεύω ψηφοφοριών. Παράγραφος 1, νέα, τροπολογία 51, υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική τροπολογία 2. Α, έφτασε η κυρία Ματσόνη. θα υποφέρετε. Συνεχίζετε με μένα. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. 59, 59, συγγνώμη, τροπολογία 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 71, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 72 που έχουμε χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Υπέρ. Με συγχωρείτε. Έχουμε χωριστή ψηφοφορία στην τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 99 υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε, ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος 99. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Λοιπόν, να σε παληθεύσουμε ηλεκτρονικά, σας παρακαλώ. Τροπολογία 100. Άρτη ψηφοφορία. Και δεν λειτουργεί στο σύστημα. Άρτη ψηφοφορία, λοιπόν. Και όντω λειτουργεί το σύστημα. Τουλάχιστον το δικό μου. Α, δεν, δεν λειτουργεί. Κάτι δεν λειτουργεί με τα μηχανήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Ονομαστική ψηφοφορία, συμφωνείτε. Δεν λειτουργεί. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ψηφίζουμε για τροπολογία 100 υπέρ. κατά Απορρίπτεται, λέει η πρόεδρος. Συγγνώμη, διορθώνει η πρόεδρος, εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αποχές, με συγχωρείτε. Έχει διαγραφεί η 102. Μάλλον πρέπει να την ψηφίσουμε, με συγχωρείτε. Υπέρ για την 102. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 104. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία 110. Περνάμε στην τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Μου λένε ότι εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Περνάμε στην 36. Χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να επαληθεύσουμε. Δεν ξέρω αν λειτουργεί τώρα το σύστημα. Όχι, δεν λειτουργεί, επομένω θα μετρήσουμε. Τροπολογία 38, ποιοι είναι υπέρ. Εννέα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 και 42 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίνεται συγχαρητήρια. Μία αποχή, συγγνώμη. Κυρία Ματσόν, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Uh, Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τη συνεργασία τους για την έκθεση αυτή και για την ψηφοφορία και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τη Γραμματεία για την πολλή δουλειά που έκανε, ιδίω η Κάρελ. Και μου αρέσουν και τα χρωματάκια στον κατάλογο ψηφοφοριών, διότι είναι πολύ χρήσιμο και ακόμα και ο κύριο Κάσμαν θα το βρει ωραίο. Έχει καιρό. Σε ευχαριστώ όλους για το ε, επιτυχές αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσίτσεστερ. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Βαλέαν είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησης, δεν είναι εδώ στην αίθουσα. Θα ξεκινήσει απευθείας λοιπόν η ψηφοφορία. Τροπολογία 1 της κυρίας Βαλέαν, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, Μπέκερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, Βάλεαν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Βάλεαν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15, Μπέκερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, η Μαϊγέρ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να κάνουμε μια παλήθευση. Υπέρ, σηκώστε ξανά τα χέρια σας. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Μέγερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Μπασέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Βαλέσα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 Βαλέσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 Βάλεαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 Μέγερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 Μπασέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 ε, έχει και προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος αντίθετος στην προφορική τροπολογία. Όχι, επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 25 ως τροποποιήθηκε από την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 Μπασέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 Βάλεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 Μπασέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 Βάλεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 Μπασέσκου υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, Baker, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, Τζανόκα, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 39, Βαλέσα, με προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αντίθετος στην προφορική τροπολογία. Ωραία, ψηφίζεται ως τροποποιήθηκε την 39 Βαλέσα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 Κάσμαν και αυτή με προφορική τροπολογία είναι κάποιος αντίθετος, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 32 του κυρίου Κάσμαν, ως τροποποιήθηκε από την προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 Βαλέσα, συγγνώμη, καταπίπτει και 34 καταπίπτει, 35 Βασέσκου υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 αν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 αν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 αν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 Κάσμαν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 37 αποσύρθηκε. Τροπολογία 40 Βαλέσα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 Νεντελτσέβα υπέρ. Κατά. Να κάνουμε μια επαλήθευση για την 38. Ε, σηκώστε και πάλι τα χέρια σας υπέρ. Ναι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 41 Μπασέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 Βάλαν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 Μπασέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 Τζανόκα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 Μπασέσκου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 Baker υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 12 βάλεαν υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 46 καταπίπτει, 47 κάσμαν υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 13 καταπίπτει, η τροπολογία 48 Κάσμαν με προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος αντίθετος στην προφορική τροπολογία, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 48 Κάσμαν ως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους. Συγχαρητήρια στη κύρια Βαλέν. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη γνωμοδότηση, στην ημερήσια διάταξη. Συντάκτρια και πάλι κυρία Βάλεαν, η οποία απουσιάζει. Αρχίζει λοιπόν απευθεία η ψηφοφορία. Τροπολογία 1 της κυρίας Νεντελτσέβα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της κυρίας Γκόντς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 μπάγκο. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, γκόνς, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8, Άουκεν Τζανόκα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Συγγνώμη, τροπολογία 15, Άουκεν κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 Γκέριγκερ Όντεμπερκ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπο... Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 Βαλέσα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 Μέγερ υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 23 για υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 μπαγκό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 γκέοντς με προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος αντίθετος στην προφορική τροπολογία. Ωραία, ψηφίζουμε την τροπολογία 25 ως τροποποιήθηκε υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 26 Κάσμαν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 27 Άουκεν Τζανόκα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31 Νεδελτσέβα υπέρ, κατά αποχές να κάνουμε μια επαλήθευση επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για την 31 Νεντελτσέβα υπέρ κατά 8 κατά, 11 υπέρ, εγκρίνεται η τροπολογία. 32 μπαγκό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 γιάρ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 πίπτη, 35 νεντελτσέβα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 για repair, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 Baker repair, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 Auken υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 Baker υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οι 40 και 41 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Abbiamo quindi chiuso la, eh, il punto relativo. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το σημείο για τις ψηφοφορίες για τα έγγραφα και τώρα θα περάσουμε στα σημεία 7 και 8 που αφορούν την έγκριση των εκθέσεων για τις διερευνητικές επισκέψεις μας. Ζητώ συγγνώμη κατόπιν υπόδειξης της γραμματείας ε, θα σας ε, πω ακριβώς τι συμβαίνει. Ε, Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μας Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την άποψη ότι ο συντονιστής της Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας έχει αναφέρει σε σχέση με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για την έκθεση όσον αφορά την επίσκεψη στη Γερμανία που αφορά επίσης και τη διαρευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία ως θέμα. Νομίζω είναι θεμελιώδους σημασίας για τις επιτυχείς δραστηριότητες της κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής ο εισηγητής από κοινού με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να καταλήξουν σε μια συμφωνία, ώστε η έκθεση που θα υποβληθεί να εκφράζει πραγματικά στο τέλος τέλος μια σφαιρική πολιτική υποστήριξη και τοποθέτηση. Θέλω να αναφερθώ στην εξαιρετική δουλειά που έγινε σε σχέση με την Ρουμανία. Αρχικά είχαμε διαφορές, σημαντικές διαφορές. Όμως, με βάση τις καλές προθέσεις του εισηγητή και των συναδέλφων, καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική λύση στο Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα εδώ και η ουσία είναι η ικανότητα να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Εκπλήσωμε κάπως από το γεγονός ότι το ΕΛΚ έχει απέναντι μια κατάσταση όπου ένα μέλος του ΕΛΚ Υποβάλλει, καταθέτει μια τροπολογία κατά της κομματικής γραμμής του ΕΛΚ και από την άλλη πλευρά, μια και θέλουμε να προλάβουμε μια τέτοια κατάσταση να επανασυμβεί στο μέλλον και εγώ προσωπικά θα καταψηφίσω όλες τις τροπολογίες πρέπει να πω που θα κατατεθούν και κατατίθενται με αυτόν τον τρόπο, διότι αντιβαίνουν το πνεύμα αυτή τη προσέγγιση σε σχέση με τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή και που πρέπει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα κιόλα και των συντακτών αναφορών. Από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρχει και μια ατμόσφαιρα, ένα περίγυρο αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν θέλουμε να έχουμε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις σε σχέση με διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες ή συγκρούσεις ιδεολογικέ. Και ως προς αυτό πάλι θα καταψηφίσω τις τροπολογίες σε σχέση με την έκθεση για την επίσκεψη την αποστολή στη Ρουμανία. Η καλύτερη λύση, πιστεύω, για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης είναι να υποβάλουμε μια έκθεση εδώ που θα αντανακλά τους λογικούς και συνετούς συμβιβασμούς που εκφράζουν όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Μπουλάν. Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να αξιολογήσω το πώς θα εξελιχθεί η ψηφοφορία όσον αφορά πάντως το ΕΛΚ. Πρέπει να σας πω ότι έκανα κάποιες προτάσεις οι οποίες ουσιαστικά συνάδουν με τα όσα είπαν και οι συντονιστές από την πλευρά των σοσιαλιστών. Είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε μία κατασυνείδηση ψηφοφορία, ελεύθερη ψηφοφορία. Εμείς σεβόμαστε τη στάση των σοσιαλιστών. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει και με τη στάση του ΕΛΚ. Οι δικές μου προτάσεις θεωρώ ότι είναι σχετικά μετριοπαθείς και τα όσα θα ψηφίσουμε δεν είναι νομοθετικό κείμενο, είναι απλώς συστάσεις συστάσεις τις οποίες υποβάλλουμε. Επομένως θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις πιστεύω. Και θα θέλω επίσης να σας πω ότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίγον να εγκρίνουμε μια, ένα κανονισμό όσον αφορά τα fact-finding missions. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεχημένα και αόριστα αυτή τη στιγμή και δεν μας επιτρέπει η σύγχυση αυτή, η ασάφεια αυτή, να καταφέρουμε να τοποθετηθούμε σωστά στη μία ή την άλλη πολιτική ομάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προτάσεις που υπέβαλα γίνονται στα πλαίσια ενός πνεύματος συμβιβαστικού, αντίθετα με τα όσα υπόθηκαν, και στις συστάσεις μου, στις συστάσεις μου λέω ότι ε, τα μέλη τα οποία συμμετέχουν στις αντιπροσωπείες αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μία επικρατέστερη θέση στη συνέχεια στα συμπεράσματα και στις συστάσεις των αποστολών αυτών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ομιλώ και τονίζω ως εισηγήτρια για την γνωμοδότηση του κυρίου Μποστινάρου από την ε, σοσιαλιστική ομάδα που δεν είχε γνωστοποίησει κάποια θέματα σε μένα. Ο τρόπος συμφωνίας μεταξύ των συντονιστών δεν συνεπάγεται κάποια υποχρέωση για τον εισηγητή να, στο να εκφράσει εκείνος ε, τις απόψεις του. Το γεγονός ότι υπάρχουν τροπολογίες είναι θετικό. Καταδεικνύει ότι η αποστολή μας με δημοκρατικό χαρακτήρα, όπου κάθε ένας είναι ελεύθερος να εκφράζει τις απόψεις του για διατάξεις, προβλέψεις κτλ. Όμως το να απαλληφθούν προτάσεις που γίνονται από συναδέρφους σημαίνει υπονόμευση. Καταστροφή και υπονόμευση του έργου που επετελέστηκε επί πάνω από ένα εξάμεινο. Συμφωνώ από την άλλη πλευρά ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες για μας σε σχέση με την αποστολή, πώς θα έπρεπε να εργαστούμε. στην σημαντική πίεση ως εισηγήτρια. Θέλω να ευχαριστήσω για το επικοδομητικό πνεύμα των εισηγητών, διότι έγιναν θετικά πράγματα. Αφήνω σε εσά να κρίνετε, συνάδελφοι, σε σχέση με τη συνείδησή σας διότι αυτή είναι η ευθύνη μας ενώπιον των πολιτών που μας εξέλεξαν. Ευχαριστώ. Ε, Κατανοώ κύριε Μποστινάρ ότι θα θέλατε εκθέσεις χωρίς τροπολογίες. Αυτό είναι η επινόηση ότι θα πρέπει να έχουμε εκθέσεις μόνο χωρίς τροπολογίες επαρτών ή θα έπρεπε να καταψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες. Συνήθως είχαμε εκθέσεις, είχαμε τροπολογίες και ψηφίζαμε υπέρ ή κατά. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίζουμε τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιώτοβα. Είχαμε μεγάλη συνένεση. Παρότι προερχόμαστε από διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες, εξετάσαμε από κοινού τις τροπολογίες. Και τώρα εδώ σε σχέση με αυτές αυτό το πρόβλημα αυτών των τροπολογιών έχουμε και δικές μου τροπολογίες και άλλων συναδέφων, άλλων πολιτικών ομάδων. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να αντιμετωπίζονται σε, από κοινού σε ένα καλάθι ισοπεδωτικά. Και πάλι σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας κυρία Γιώτο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν γνωρίζω απόλυτα τις λεπτομέρειες σε σχέση με την αποστολή διακρύβωσης στο Βερολίνο, αλλά ξέρω τι συνέβη στη Ρουμανία. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Μποστινάρου, θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι η δίκη του κυρίου Μποστινάρου ή των σοσιαλιστών σε σχέση με αυτά τα θέματα. Είναι μάλλον μια ριζοσπαστική αλλαγή θέσης του συναδέλφου και καθώς άλλαξε το καθεστώς η κυβέρνηση στη Ρουμανία, πολύ καλά γνωρίζετε ότι ο κύριος Μποστινάρου προσπαθούσε να ασκήσει πίεση στους συναδέφους για κάποιες ετροπολογίες και για την εισαγωγή σε αυτή την έκθεση κάποιων στοιχείων που δεν ανήκουν σε αυτή την έκθεση. Αυτό είναι κάποια τελείως διαφορετική λοιπόν προσέγγιση, τελείως διαφορετική ιδέα. Τον άρχεται κάποιος εδώ και να λέει ότι δεν είναι θεμητό και δεν είναι συνετό για κάποιους συναδέλφους να, να καταθέτουν τροπολογίες αυτό δεν είναι θετικό σε σχέση με τοποθέτηση Ευρωβουλευτή. Νομίζω έχει δικαίωμα ο συνάδελφος να καταθέσει όποιες τροπολογίες επιθυμεί. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορούν να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν. Αλλά θέλω να αποσαφηνίσω το γεγονός ότι αυτή η τοποθέτηση οφείλεται στο ότι ο κύριος Μποστινάρου είχε μία διαφορετική αντιφατική άποψη σε σχέση με στοιχεία για την έκθεση στη, για τη Ρουμανία. Τώρα δεν προσπάθησε να εξεύρει μια συνενετική λύση. Τώρα έχει, έχουν την εξουσία στη Ρουμανία και έτσι περιπλέκεται το θέμα. Yes. Εντάξει κύριε Βίλαντ, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ζητώ να μην ξανανοίξουμε και πάλι μια συζήτηση, εντάξει. άρχισε η ψήφιση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση και να την ξαναξεκινήσουμε για αυτό το θέμα. Βρισκόμαστε στο τέλος του κοινοβουλευτικού μας έργου πριν από τις διακοπές. Είναι η τελευταία μας συνεδρίαση. Θα σας ξαναδώσω τον λόγο μετά, τον κύριο Βίλαν, μετά από τον κύριο Βίλαντ και έτσι μπορείτε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση για δύο λεπτά. Ο κύριος Βίλαντ πρώτος παρακαλώ. Ζήτησα τον λόγο για διαδικαστικό και θα ήθελα επ' αυτού να τοποθετηθώ. Πρέπει να ψηφίσουμε νομίζω τώρα. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Και όλα αυτά τα γεγονότα δείχνουν με σαφήνεια ότι η δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή, και θέλω να το ζητήσω αυτό, στη συνέχεια για, την, για τις fact-finding missions και τα follow-ups για τις αποστολές μας, διακριβωτικές αποστολές, πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες που θα ισχύουν. Δεύτερον, για την διακριβωτική αποστολή στο Βερολίνο πρέπει να πω ότι η πρόεδρος της Επιτροπής είχε πει πιο πριν ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τροπολογίες στα συμπεράσματα. Εγώ στη συνέχεια τις δικές μου τροπολογίες για τα συμπεράσματα τις απέσυρα. Τρεις τροπολογίες ε, που ε, καταλήγουν τώρα σε ψήφιση, θεωρώ ότι είναι αθέμητες αυτές οι τροπολογίες. Δεν μπορούν να είναι αποδεκτές. Μόνο δύο λόγια, κύριε Μποστινάρου. Δύο λόγια μόνο. Κατανοώ απόλυτα ότι ο αγαπητός Ρουμάνος συνάδελφος κύριος Λουχάν, επειδή ποτέ δεν συμμετείχε στην αντίστοιχη Κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν γνωρίζει τους κανονισμούς και τις διατάξεις. Μπορείτε να είσαστε εσείς μάρτυρας, κυρία Ματσόνη, για την ποιότητα της δουλειάς που κάναμε από κοινού. Και τέλος, γιατί αν ο ε, ο συντονιστής του ΕΛΚ, δεν είναι ικανοποιημένος ή είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο με τον οποίο οι τροπολογίες κατατέθηκαν από κάποιους από τους δικούς του συναδέλφους, γιατί να κατηγορεί τους ασυρδημοκράτες για αυτά τα προβλήματα που έχει το ΕΛΚ, το ίδιο το ΕΛΚ. Δικό μου συμπέρασμα είναι να συνεργαστούμε καλύτερα με λογικό τρόπο για να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή για μένα. Πρόεδρος, παρακαλώ συνάδελφοι. Τώρα, ε, κοιτάξτε. Σας έδωσα το λόγο διότι είχα θεωρήσει ότι έπρεπε ο καθής να έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, τη θέση του. μετά από πολύ σοβαρή δέσμευση της Επιτροπής μας ε, προκειμένου να εγκρίνουμε όχι μόνο την έκθεση για την ε, ε, διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο αλλά και αυτή στη Ρουμανία. Βεβαίως η ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από το κοινό πνεύμα το οποίο προσπαθούμε ε, να, επιδείξουμε ενώπιον των πολιτών γιατί βασικά αυτή θα έπρεπε να είναι η δουλειά μας, να στεκόμαστε πλάι στους πολίτες μας. Ε, είναι ακόμα ελπίδα αυτό κύριε Μποστινάρου, δεν έχει πραγματοποιηθεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή να είμαστε πραγματικά υπεράνω πολιτικών κομμάτων και να προωθούμε τις αρχές της δημοκρατίας εάν αρχίσουμε να κάνουμε εξαιρέσεις στους κανόνες. Κάποιος το πρότεινε, εγώ ως πρόεδρος ε, δέχομαι τις προτάσεις από όλες τις πολιτικές ομάδες και από εκεί και πέρα τις συζητούμε. Ε, προσωπικώς δεν συμφωνώ με την άποψη να αλλάζουμε κανόνες ε, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διεξάγεται μια αποστολή και από εκεί και πέρα πώς θα συντάσσεται η έκθεση που πρέπει να γίνεται στη συνέχεια της και δεν νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τον αντικειμενικό μας σκοπό. Η κατάθεση τροπολογιών, όσο και αν θεωρείται λογική ή μη ανάλογα με το πώς το αντιμετωπίζει ο καθένας, ούτως ή άλλως είναι δυνατή για οποιοδήποτε έγγραφο συζητούμε εδώ στην Επιτροπή, διότι είναι η αρχή που ε, διέπει και σε αυτή την περίπτωση της εργασίας μας, δηλαδή της δημοκρατίας. Εάν κάποιος διαφωνεί, ούτω ή άλλω ε, η Επιτροπή είναι αυτή η οποία έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να αποφασίσει. Ψηφίζουμε λοιπόν για να καταλήξουμε στην κοινή θέση, τη θέση της πλειοψηφίας, σαφώς δεν είναι ομόφωνη θέση, του οργανισμού που εκπροσωπούμε μεμονωμένα αλλά και συλλογικά όλοι μας. Μπορούμε να εκφράσουμε μια πολιτική αντίθεση για κάποιον ε, ο οποίος ε, είχε συνεκτική στάση ή δεν είχε συνεκτική στάση, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε αντίθετοι στο να μπορεί ο καθής να κατεθέσει την τροπολογία του και να την απορρίψουν ή να την εγκρίνουν τα μέλη της Επιτροπής μας. Σας παρακαλώ λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τώρα την ε, ψηφοφορία για την πρώτη έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη ε, στο Βερολίνο, ε, η οποία έγινε σχεδόν πριν από ένα χρόνο και το επισημαίνω αυτό. Η κεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν η κυρία Ιώτοβα και επομένως αυτή ήταν και η αρμόδια να συντονίσει τις εργασίες για την εκπόνηση της έκθεσης Παρουσιάστηκαν κάποιες τροπολογίες, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Τροπολογία Μπουλάν, υπαριθμόν 1. Άρχεται η ψηφοφορία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, διότι... Ε, δεν κατάλαβα με τον τρόπο που σηκώσατε τα χέρια σας ποιος ψήφιζε τι υπέρ. Κατά. 9 κατά, 8 υπέρ, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 μπουλάντ, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 μπουλάν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. sull'emendamento Για την τροπολογία 4. Συγγνώμη, δεν αφορά την τροπολογία 4. Έχει προταθεί. Ε, κύριε Μπουλά, μισό λεπτό να ολοκληρώσω μπορείτε να είστε αντίθετο στην προφορική τροπολογία. λεμένταμεν. Αποσύρθηκε η προφορική τροπολογία. Όχι προφορική τροποποίηση, αλλά η τροποποίηση, η τροπολογία όπως έχει τυπωθεί στο έγγραφο, όπως είναι τυπωμένο. Ωραία, προχωρούμε λοιπόν με την ψηφοφορία τροπολογία 4. Γιάρ Βίλαντ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ξαναψηφίσουμε την 4 υπέρ. Κατά. Εννέα υπέρ. 8 κατά, εγκρίνεται. Η ε, διαδικαστικό, κύριε Μπουλάν, διότι είμαστε μέσω ψηφοφορία. Ψηφίζουμε, κύριε Μπουλάν. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε συζήτηση. Μα δεν ανοίγω συζήτηση να σας ζητήσω κάτι. Δεν είμαι πεπισμένος, δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα της προφορίας για την τροπολογία υπαριθμών 1. Νομίζω ότι δεν έγινε σωστός υπολογισμός, δεν έγινε σωστή καταμέτρηση των ψήφων. doesn't, uh, it work. Ναι, αλλά δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορείτε να ελέγξετε αν μπορεί να λειτουργήσει το μηχάνημα. Έχει ζητηθεί επαλήθευση, δυστυχώς όμως πρέπει να γίνει διανατάσεως χειρός, διότι δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Ο κύριος Μπουλάν έχει ζητήσει επαλήθευση για την ε, τροπολογία 1, έτσι. Ο κύριος Μποστινάρο, κοιτάξτε να δείτε, ε, με τη συζήτηση χάνουμε ε, τη χρόνο. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε στην 1. Έχουμε ψηφίσει 2, 3 και 4 και ξαναγυρνάμε στην 1. Ε, ψηφίστηκε. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες. Συγγνώμη, είμαι αντίθετο. Η πρόεδρος. Δεν ε, αλλάζουμε τους κανόνες. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε μια δεύτερη καταμέτρηση υπήρξε κάποιο πρόβλημα διότι ο κύριος Μπουλάν ζητούσε το λόγο και εγώ νόμιζα ότι ήθελε να λάβει το λόγο για να ξανασυζητήσουμε το ζήτημα και στην πραγματικότητα ήθελε το λόγο απλώς και μόνο για να γίνει μια επανάληψη της καταμέτρησης. Εκτός μικροφώνου του κύριου, το σχόλιο του κύριου Μποστινάρου. Τροπολογία 1, σας παρακαλώ. Να κάνουμε έναν έλεγχο. Who is for? Υπέρ. Eight. In favor. Οκτώ υπέρ. Oh. Frau Vorsitzende. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, για διαδικαστικό. Συγγνώμη κύριε Βόλε, ε, Βίλαντ, υπάρχει πρόβλημα με το μηχάνημα και δυστυχώς πρέπει να σας υποχρεώνω κάθε φορά να ε, καταμετρήσει για να είμαστε βέβαιοι. Κύριε Βίλαντ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, για διαδικαστικό πρώτον, η τροπολογία μετρήθηκε πιο πριν και είχαμε αποτέλεσμα. Δεύτερον, ο συνάδελφος Μποστινάρο έχει δίκιο δεν μπορεί να πάμε πίσω ως κοινοβούλιο επειδή κάποιοι δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία ή έρχονται άλλοι καινούργοι. Αυτό είναι ακριβώς τον λόγο γιατί οι ψηφοφορίες άμεσα ελέγχονται, καταμετρώνται ή ε, υιοθετείται η άποψη του Προέδρου για το αποτέλεσμα. Τρίτον, δεν είδα σε καμιά κοινοβουλευτική επιτροπή παρατηρήσεις από τους συμβούλους ε, να ακούγονται. Αν γίνονται τέτοια πράγματα να κλείσουμε το μαγαζί. Ευχαριστώ. Κύριε Βέιλαντ, επαναλαμβάνω. Ο κύριο Μπουλάν είχε ζητήσει το λόγο και εγώ δεν του τον έδωσα διότι θεώρησα ότι ζητούσε το λόγο για να ξαναξεκινήσει τη συζήτηση. Επέμεινε και μόνο μετά κατάλαβα ότι ζητούσε απλώ επαλήθευση. Θα μπορούσε να μου είχε πει τσεκ και να το είχα καταλάβει, δεν μου το είπε και υπήρξε μια παρανόηση. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να επαληθεύσουμε κατά πόσον ε, ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να χάνουμε χρόνο να το συζητάμε, διότι δεν ωφελεί κανέναν. Τώρα, αν είναι 8, 9 ή 10, μπορούμε να το επαναδειθεύσουμε σε ελάχιστο χρόνο, εάν σταματήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτή η ένσταση. Οι συνάδελφοι δεν άλλαξαν, δεν ήρθε κανεί στην αίθουσα από την ώρα που αρχίσαμε να ψηφίζουμε πριν από τρία λεπτά και επομένω η κατάσταση είναι ακριβώ η ίδια. Εάν υπήρξε λάθο από πλευρά Προεδρία ή Γραμματεία στην ε, ε, καταμέτρηση, Γι' αυτό ακριβώ το λόγο γίνεται η επαλήθευση. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο περίπλοκο. Σα παρακαλώ πολύ λοιπόν, σηκώστε τα χέρια σα και μετά από αυτό δεν δέχομαι καμία άλλη υπόδειξη από κανέναν στην αίθουσα. Ποιο είναι υπέρ λοιπόν τη τροπολογία παριθμών 1. No. No, six, seven, eight, nine. Ten. Ten. votes in favor. Chi è contrario? Εννέα λοιπόν υπέρ. Ποιος είναι κατά? Otto contrari. Κύριε Πρόεδρε. Remind Ο κύριο Μποστινάρου διακόπτη. Κυρία Πρόεδρε, κάποια στιγμή όταν συζητούσαμε το θέμα των μέσων μαζική ενημέρωση στη Ρουμανία, είπατε ότι οι κανόνε ισχύουν μόνο για την Επιτροπή και άπαξ και έχει ε, περάσει το ζήτημα, κανένα δεν μπορεί να αμφισβητήσει την, ε, το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Αυτό είναι βάση κανόνων. Και η διάσκεψη των Προέδρων τότε αποφάσισε να επανοργανώσει την ψηφοφορία γνωρίζετε την ιστορία τώρα, δεν χρειάζεται να επεκταθώ περαιτέρω επί του ζητήματος. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ξαναψηφίζουμε και να επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία εφόσον έχει γίνει η ψηφοφορία και έχει περάσει, από η τροπολογία. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιο στην αίθουσα και να μπαίνει και να βγαίνει γιατί αλλάζει η κατάσταση ο κύριος Βαλέσα είναι ο αναπληρωτής συντονιστής του ΕΛΚ. Θα ήθελα να μας πει και αυτό στην άποψή του. Μπορεί το ΕΛΚ λοιπόν να αντιδράσει και να δεχτεί αυτή την κατάφορη παραβίαση των κανόνων μας. Σας παρακαλώ να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία σε άλλε επιτροπέ. Η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα, ο κύριο Μποστινάρου εκτό μικροφώνου. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εφεύρουμε κάτι καινούριο, κύριε Μποστινάρου. Και μάλιστα εγώ είμαι υπεύθυνη για την προεδρία της Επιτροπής αυτής και αναλαμβάνω λοιπόν εγώ ίδια προσωπικά την ευθύνη για το τι έχουμε πράξει. Νομίζω πάντως ότι για κάθε ψηφοφορία οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει επαλήθευση. Επαληθεύσαμε λοιπόν την ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη τροπολογία και μεταξύ των δύο ψηφοφοριών, της πρώτης δηλαδή και της επανάληψής της, τίποτα δεν άλλαξε όσον αφορά τη σύνθεση της αίθουσας. Σας το εγγυώμαι. Ο συνολικός αριθμός παραμένει ο ίδιος. Δεν τροποποιήθηκε η σύνθεση της αίθουσας. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργούν τα μηχανήματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τώρα λειτουργούν, μου λένε, αλλά δεν μπορούμε να επαναλάβουμε εκ νέου την ψηφοφορία. Για τις επόμενες ψηφοφορίες θα χρησιμοποιήσουμε πάντως συσκευές μας. Δεν νομίζω πάντως ότι αποτύχαμε κατά την εφαρμογή των κανόνων. Και νομίζω ότι θα πρέπει κάθε φορά να προσπαθούμε να βλέπουμε ποια είναι η πραγματική τοποθέτηση της Επιτροπής. Και αν η Επιτροπή ψηφίζει 9 υπέρ 8 κατά, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε το αποτέλεσμα αυτό. και δεν πρόκειται να επανέλθω να αναθεωρήσω το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών μας, εκτός και αν οι συνάδελφοι μου ζητήσουν επαλήθευση αμέσως μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Θα πρέπει να μου λέτε ζητώ επαλήθευση και όχι απλώς ζητώ το λόγο, εντάξει. Mr. Wieland. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. <clears throat> κυρία Πρόεδρε. Τώρα δεν βοηθάει, δεν βοηθάει όταν επαναλαμβάνουμε τις θέσεις ο ένας και ο άλλος. Είπατε επομίζεστε την ευθύνη, ευθύνη γι' αυτό. Θέλω να πω με σαφήνεια ότι άλλαξαν συνάδελφοι άποψη και γι' αυτό μια τέτοια διαδικασία ούτε στην Ολομέλεια ούτε σε άλλες κοινοβουλευτικές ήθιστε να ακολουθείτε. Όταν λέτε εσείς επομίζεστε την ευθύνη, εγώ θέλω ρητά στα πρακτικά να καταχωρηθεί η διαμαρτυρία μου γι' αυτό. Ε, Σαφέστατα θα ληφθεί υπόψη, κατά γράμμα, θα ζητήσω από τη γραμματεία να ε, περάσει τα πρακτικά. Συνεχίσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Ο κύριος Μποστινάρου. Χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για την ε, νέα καταμέτρηση και θα ήθελα επίσης να ζητήσω να εξετάσουμε κατά πόσον εφαρμόστηκαν καταλήλω οι κανόνε στη διάρκεια τη ψηφοφορία, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Έχετε κάθε δικαίωμα να τους δείστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες επαλήθευσης που έχετε στη διάθεσή σας και αν ε, οι ανώτεροι μας αποφασίσουν ότι έσφαλα θα δεχτώ και θα διορθώσουμε την κατάσταση. Συνεχίζουμε η τροπολογία 5 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 4, τροπολογία 6, Γιάρ Βίλαντ, υπέρ. Κατά. Άποχες. Σας παρακαλώ, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, ώστε να μην χάνουμε χρόνο, διότι μου λένε ότι τώρα λειτουργούν τα μηχανήματα. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, λοιπόν, από εδώ και πέρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 6 Γιαρ Βίλαντ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiudiamo la votazione. Πέραση ψηφοφορία. L'emendamento Απορρίπτεται 10 ψήφοι κατά, 8 υπέρ. Τροπολογία 7, Μπουλάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία από εδώ και πέρα. Πέραση ψηφοφορίας. 10 υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 8 μπουλά. Ε, la votazione. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Dieci favorevoli, 8 contro. 10 υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία κολάρκα Καβομπίνσκα καταπίπτει. Τροπολογία 9 Τζανόκα. Άρχεται η ψηφοφορία. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Έχω διαρκώς προβλήματα με, το, με τη συσκευή εδώ μπροστά. Allora, riapriamo la votazione sulle... Ψηφίζουμε και πάλι λοιπόν. Τροπολογία 9, Τζανόκα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. 17 υπέρ, 1 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 11, Μπουλάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 16 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 μπουλάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 1 κατά. Τροπολογία 14, Μπουλάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 13 μπουλάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκαέξι υπέρ, ένας κατά. Τροπολογία 14 μπουλάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 1 κατά. Η 15 καταπίπτει. Η 16 Τζανόκα. άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 17 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 Μπουλάν. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 15 υπέρ, ένας κατά, δύο αποχές. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, ένας κατά. Καταπίπτουν οι 19 και 21. Τροπολογία 20 μπουλάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 17 υπέρ. Τροπολογία 25. Πανομοιότυπη με την 20, ταυτόσημη. Εγκρίνεται λοιπόν γιατί ήταν ταυτόσημη με την 20, εγκρίνεται και 25. Τροπολογία 22 μπουλάν. Πέρας ψηφοφορίας. 10 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23, Γιάρ Βίλαντ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 10 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία. Καταπίπτει η 24. Τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 11 υπέρ, 6 κατά. Τροπολογία 27, μπουλά, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 8 υπέρ, 10 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28, Μπουλάν. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 11 υπέρ, 6 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 29, Μπουλάν. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 1 κατά, 2 αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, Μπουλάν. άρτε ψηφοφορία. Πέρας. 7 υπέρ, 9 κατά, μία αποχή, απορρίπτεται. Τροπολογία 31, Μπουλάν. άρτε ψηφοφορία. Πέρας. 10 υπέρ, 7 κατά, η τροπολογία εγκρίνεται. Τροπολογία 32 του κ. Μπουλά. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. 16 υπέρ. Μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 Μπουλά. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. 8 υπέρ. 7 κατά. 2 αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 Μπουλά. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. 7 υπέρ, 8 κατά, 2 αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Μπουλάν. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση με 11 ψήφους υπέρ, 6 κατά και μία αποχή. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για να αποφύγουμε παληθεύσεις, ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις τρεις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Αν δεν έχετε λοιπόν αντίρρηση... Άρχεται η ψηφοφορία για τις α, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για την έκθεση αυτή. Αναφερόμαστε πάντα στη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία. Τροπολογία υπαριθμών 1. Πρέντα Μπασέσκου, άρτη ψηφοφορία. Άρτη ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 1. Πέρας. 7 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Πρέντα Μπαζέσκου. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας ένας υπέρ, επτά ψήφοι κατά, έξι αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 3, πρέντα μπαζέσκου, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Μία ψήφο υπέρ, επτά ψήφοι κατά και 7 αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση το σύνολο της έκθεσης, άρτη ψηφοφορία, πέρας, 10 ψήφοι υπέρ, 4 αποχές, εγκρίνεται η έκθεση. 10 ψήφοι υπέρ, 4 αποχές. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ψηφοφορία πλέον. Παρακαλώ συνάδελφοι να ξεκινήσουμε τώρα με το επόμενο σημείο. στην ημερήσια διάταξη στο σημείο υπαριθμών 9 έχουμε την ετέσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του 2011, ε, την οποία έχω αναλάβει εγώ. Είμαι η συγγήτρια. Κύριε Ποστονάρου, σας παρακαλώ. Υπάρχει ένα σχέδιο έκθεσης, ε, το οποίο στην ε, προηγούμενη συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου συζητήθηκε και με, είχαμε παρουσία του Ευρωπαίου Δημοσιολαβητή, ο οποίος μας μίλησε για την έκθεση του για το 2011. Σας παρουσιάστηκε αρκετά δεξιοδικά εδώ στην Επιτροπή μας. Έχουμε τα στοιχεία της δραστηριότητας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Και προς αυτό κάνουμε μια έκθεση κάθε χρόνο. Τα στοιχεία που έχουμε για το 2011 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ε, σίγουρα θετικά δεδομένων και των ε, απαιτήσεων που έχουμε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Γνωρίζουμε ότι ο Ευρωπαίος ε, Διαμεσολαβητής συμμετέχει στο δίκτυο Ευρωπαίων πολιτών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την ε, φροντίδα των Ευρωπαίων πολιτών και την προστασία τους. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε κάποια στοιχεία που μας δείχνουν ότι έχουμε αύξηση του αριθμού των αναφορών που κατατέθησαν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και που επιλήθηκαν με αποτελεσματικό τρόπο. Έχει υπάρξει και συνολική αύξηση των αριθμό των αναφορών που κατατέθησαν προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όπου υπήρχαν εσφάλματα. Ε, αυτά ε, καταδεικνύουν ότι ε, είναι σίγουρα θετική η έκβαση. Το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των διαδικασιών Στη διάρκεια του έτους που μετά από τις αναφορές ε, προχώρησαν από τον ίδιο το διαμεσολαβητή σημαίνει ότι βελτιώνεται η ε, ίδια η δομή του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι υπάρχει μείωση των αναφορών προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λιγότερες δηλαδή αναφορές που αφορούν ε, ε, εσφαλμένη ε, διαχείριση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γεγονός ότι μειώθηκε ο αριθμός των αναφορών αυτών θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυξήθηκε ο αριθμός των αναφορών Ε, καταγγέλουν τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως ε, επιδείνωση της ε, διαχείρισης των υποθέσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο. Είναι αυτή που εκτελεί όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι φυσικό να είναι ε, το θεσμικό όργανο προς το οποίο απευθύνουν ε, ε τις περισσότερες καταγγελίες τους ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και αυτό αναφέρεται στο σημείο 19. όπου εκεί αναφέρεται και το πόσο καλό αποτέλεσμα είχαμε στις δραστηριότητες ε, του 2011 από το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, διότι χρησιμοποιούνται συστήματα ε, πληροφορικής και επικοινωνίας με τους πολίτες ε, πολύ πιο προηγμένα από ό,τι στο παρελθόν. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαθέτει πλέον ένα εγχειρίδιο για τις καταγγελίες προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, διαθέτει ένα σύστημα πληροφορικής μέσω διαδικτύου πάρα πολύ προηγμένο και φυσικά αυτό οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα για την ε, ε, προηγούμενη χρονιά. Έχουμε κάποια αναλυτικά στοιχεία στην έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή από αυτού και ε, εγώ έχω αναφέρει στην έκθεσή μου μόνο εν είδη παραδείγματος κάποια. Η πρόταση λοιπόν που κάνω στην έκθεσή μου είναι να στηρίξουμε τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στη διάρκεια του 2011. Καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν όλα τα ε, ε, τα όργανα του δικτύου ε, προς τους πολίτες ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικά είναι τα καθήκοντα τα οποία διεξάγουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε ιδιαίτερα να προωθήσουμε την συμμετοχή των πολιτών και να προχωρήσουμε ε, να προχωρά συνεχώς η δημοκρατία. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Θα ήθελα να ακούσω υποδείξεις και προτάσεις των συναδέλφων, εάν υπάρχουν. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Άου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα... Συγγνώμη να περιμένω μια στιγμή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενέσω αυτή την έκθεση. Είναι εξαιρετική και με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι υπάρχει άμεση αναφορά σε βελτιώσεις όσον αφορά την διοίκηση και όσον αφορά την εξυπηρέτηση, την τα συμφέροντα του πολίτη που θα βρίσκονται πάνω-πάνω σε σχέση με τις υπηρεσίες, τις διοικητικές υπηρεσίες. Αυτό είναι σημαντική πρόοδος. Είναι κάτι το κοινό για όλους. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να κατανοήσει η διοίκηση αυτό το σημείο, ή πάλι και ελπίζω ότι κάποτε θα το κατανοήσουν και εκείνοι απόλυτα. Ένα πράγμα που θα ήθελα να εκφράσω με απόλυτη σαφήνεια. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από μια συγκεκριμένη χώρα δεν αντανακλά μια χειρότερη κατάσταση υποχρεωτικά σε σχέση με άλλες χώρες όπου υπάρχουν λιγότερα παράπονα από αυτές. Είτε υπάρχουν ιδιαίτερα ενεργοποιημένοι πολίτες που συνειδητοποιούν το τι μπορούν να πράξουν και έχουν εμπιστοσύνη στον διαμεσολαβητή και έτσι απευθύνονται σε αυτόν, ή ταυτόχρονα σε άλλες χώρες που δεν υπάρχουν πολλά παράπονα, ίσως έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειές τους ε, οι πολίτες, έχουν απογοητευτεί, έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια, πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, ό,τι και να κάνουν. Λοιπόν, κάποια σχόλια απλά για το γεγονός ότι θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις και καταστάσεις που δεν αντανακλούν υποχρεωτικά τα παράπονα και οι αναφορές ε, με τα παράπονα αυτά μια αρνητική κατάσταση στην κοινωνία υποχρεωτικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χουντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, και η δική μας εκτίμηση είναι και συμφωνούμε με τα βασικά σημεία που έχετε τονίσει στην έκθεσή σας. Ε, και συνολικά έχουμε καλή γνώμη για την ε, δραστηριότητα του διαμεσολαβητή. Αυτά που αναφέρετε στην έκθεσή σας και τη βελτίωση των επιδόσεων είναι σημαντικά πράγματα έχουν συμβεί, όπως επίσης και η προσπάθεια που κάνει ο διαμεσολαβητής να αντιμετωπίσει τα αιτήματα των πολιτών, όχι ως απειλή, αλλά ως μια προσπάθεια να εξευρεθούν λύσεις σε προβλήματα που έχουν εμφανιστεί. Αν κάτι θα ήθελα να παρατηρήσω, είναι πρώτον ότι γενικώ γενικώ ε, ε, με διαβαθμίσεις βεβαίως στους Ευρωπαίους πολίτες των χωρών, ε, στους πολίτες δηλαδή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οικία η διαδικασία να παραπέμπουν παράπονά τους, αιτήματά τους προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Υπάρχει ακόμα θέμα ευρύτερης ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών ως μια δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και το δεύτερο που έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική και δεν είναι θέμα του διαμεσολαβητή, αν αυτά τα φαινόμενα που έχει την αρμοδιότητα να αντιμετωπίσει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και που άπτονται, συνδέονται με το θέμα της καλής διοίκησης, της χρηστής διοίκησης, είναι θέμα χρηστής διοίκησης ή πολιτικής που πλήττει τα συμφέροντα των πολιτών. Εκεί η πολιτική εκτίμηση δεν είναι εύκολη να γίνει και βεβαίω δεν είναι θέμα του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Αν είναι έτσι τα πράγματα και τελειώνω, η τελευταία λοιπόν λύση, στήριξη, αποσαφήνιση τέτοιων καταστάσεων που σημαίνει βοήθεια στη δουλειά του διαμεσολαβητή ή ανάθεση των ευθυνών στα πολιτικά όργανα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες ως ερετό όργανο, τις προσπάθειες του διαμεσολαβητή. Να τον περιβάλλει με την εμπιστοσύνη, κάνοντας παρατηρήσεις ε, για, τη δουλειά του, ούτως ώστε να τον βοηθήσουμε να μπορέσει να δίνει απαντήσεις, να διαμεσολαβεί, να λύνονται προβλήματα και να έχει καλύτερες επιδόσεις. Συμφωνούμε βασικά με την έκθεσή σας κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντίκε για τη δική σας τη συνεισφορά. Ε, Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει την άποψή της ε, η κυρία Κάρμεν Μπράισινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι στη συνεδρία στις 19 η Ιουνίου ήδη εξαντλητικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθετήθηκε σε σχέση με την έκθεση του διαμεσολαβητή. Δεν υπάρχει κάτι που να ήθελα να προσθέσω σήμερα ξεχωριστά. Πέρα από το γεγονός ότι καλωσορίζω τη δική σας έκθεση, υποστηρίζοντας πλήρως τα συμπεράσματά σας στην έκθεσή σας και τονίζοντα ότι κατά τη διάρκεια του έτου που καλύπτεται από αυτή την έκθεση οι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, διαμεσολαβητή εμβαθύνθηκαν, αναπτύχθηκαν σημαντικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει αυτή την θετική συνεργασία με το διαμεσολαβητή και καλωσορίζει έτσι προς αυτή την κατεύθυνση τα δικά σας συμπεράσματα στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 20 Ιουλίου Περιμένω λοιπόν ε, προτάσεις σας. Ελπίζω να έρθουν και από τους ε, απόντες συναδέλφους, ώστε να βελτιωθεί και το σχέδιο της εκθεσής μου. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα σημεία της ημερήσιας διάταξης ε, που αφορούν τη συζήτηση και μπορούμε να περάσουμε τώρα στο πρώτο σημείο στις αναφορές των πολιτών. Έχουμε λοιπόν την αναφορά 313 του 2007, την 670 του 2009 και την 58 του 2010 που αφορούν το εθνικό χρέος της Αργεντινής και την αδυναμία της χώρας να καταβάλει τα οφειλόμενα σε κατόχους ομολογιών. υπάρχουν ε, σαφείς ε, αποδείξεις από πλευράς Ευρωπαίων πολιτών, ε, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, διαθέτουν κρατικά ομέλιγα και δεν υπάρχει ιδέουσα προσοχή από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για την καταγγελία που έκαναν και υπάρχει και μια γενικότερη αδιαφορία διότι προωθούνται εμπορικές συμφωνίες άλλης φύσεως ε, με την Αργεντινή και δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταγγελίες ε, που έχουν ε, υποβάλει οι πολίτες αυτοί στις χώρες τους αλλά και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι αναφέροντες δεν είναι παρόντες, έχουν αποστείλει Ε, περαιτέρω έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή μας για να μας ενημερώσουν ε, για το θέμα. Μας έχουν δώσει και κάποια περισσότερα νέα. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι αυτές οι αναφορές ε, έχουν ήδη εξεταστεί και στο παρελθόν από την Επιτροπή μας, η οποία Επιτροπή μετά και από τη συζήτηση με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε αποφασίσει να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές αυτές προκειμένου να εξωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επενεξετάσει τη θέση της που θέλει να κλείσει τα θέματα αυτά και θεωρεί ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητά μας ε, στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε μας είχε πει ότι τα ζητήματα τα οποία θέτουν ε, οι αναφέροντες αφορούν εθνικές αρμοδιότητες και θα έπρεπε να επιληθούν ε, σε διμερές επίπεδο. Στη συνέχεια βέβαια είχαμε μία γνωστή υπόθεση ε, στην οποία εμπλέκεται εν γέννη η ισπανική οικονομία αλλά και η οικονομία άλλων χωρών εμέσως διότι ξεκίνησε η διαβόητη υπόθεση Ρέψολ, για την οποία αντίθετα με τα όσα είχαν συμβεί σε άλλες υποθέσεις που υπήρχαν σε κρεμότητα με την Αργεντινή, εκεί ε, είχαμε παρέμβαση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι τάχθηκαν υπέρ των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την ε, ε, απόφαση η οποία θεωρήθηκε ε, λανθασμένη και αντίθετη προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς της επιχείρησης που σας ανέφερα. Ε, το περιστατικό αυτό εξώθησε τους αναφέροντες λοιπόν να επισημαίνουν ότι έχει αλλάξει η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς σήμερα θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να ακούσουμε εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν όντω έχει αλλάξει στάση της, αν, αν δεν έχει αλλάξει στάση ε, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ε, συμπεριφοράς ε, των αρχών της Αργεντινής ενώπιον πολιτών μεμονωμένα και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της λανθασμένης συμπεριφοράς του κράτους της Αργεντινής ε, προς ε, ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν το λόγο ε, στην εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αλεξάνδρα Χουτουνίδης. Δώση γνώμη για τη λανθασμένη προφορά του ονόματό σας. Um, Ευχαριστώ. Γεια σας. Υπό το νόμο για τις επενδύσεις ομόλογα είναι επενδύσεις και οι κάτοχοι ομολόγων είναι επενδυτές και όσον αφορά τις τρίτες χώρες που εμπίπτουν υπό την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των αναφερόμενων, το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο είναι η διμερή συμφωνία επενδύσεων μεταξύ Αργεντινής και Ιταλίας, η διμερή σύμβαση. Οι επενδυτές όταν είχαν καταβα... υποβάλει την πρώτη αναφορά στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναφορών είχαν ήδη προσφύγει για διαιτησία υπό την ρήτρα ε, διαιτησίας που προβλεπόταν σε σχέση με αυτό το νομοθέτημα άμεσα κατά της Αργεντινής και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαιτησία το θέμα αυτό σύμφωνα με τους κανονισμούς της Σύμβασης της Washington για την διευθέτηση επενδυτικών προβλημάτων και επιμάχων σημείων όσον αφορά επενδύσεις ε, και σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ότι αυτή η σύμβαση που διέπει τις διαδικασίες διαιτησίας προβλέπει ότι ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία διαιτησίας το κράτος του επενδυτή δεν θα έπρεπε να κάνει κάποια βήματα ή διαβήματα για διπλωματική προστασία ή άλλη επέμβαση ενώ τα δικαιώματα διπλωματικής τέτοιας παρέμβασης μπορούν νόμιμα να διασφαλιστούν υστερότερα. Αυτή είναι η διαφορά με τη Repsol που σε σχέση με τα όσα γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προηγούμενη φάση είχε συμβεί αυτό όταν δεν υπήρχε το θέμα διατησίας και γι' αυτό θεωρεί σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει τις πολιτικές ανησυχίες σε σχέση με το περιθώριο το οποίο υπήρχε να υπάρξει μια φιλική συμφωνία πιο πριν και ένας φιλικός συμβιβασμός πριν από αυτή τη δράση. Ιδιαίτερα όσον αφορά την αναφορά 58, όσον αφορά την προσφορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι αυτή η προσφορά δεν υφίσταται πλέον. Συνέβη το 2010 έγινε και ως προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει απλά αυτά τα οποία ίσχυαν τότε και είχαν εκφραστεί προηγούμενα και μέσω επιστολής του Επιτρόπου Μπαρνιέ που είχε τοποθετηθεί σχετικά. Αυτή η προσφορά έγινε σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν ώστε να προστατεύεται η προστασία, να προστατεύονται τα στοιχεία που αφορούν επενδύσεις και να προστατεύονται οι επενδυτές. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ε, δεν είχα προβλέψει να κάνω παρέμβαση. Ε, είχα έρθει άλλη ερώτηση. Ελπίζω να μην σας ε, ε, δημιουργώ σύγχυση. Εάν θεωρείτε λοιπόν ότι στην παρέμβασή μου δεν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να σχολιάσετε, δεν υπάρχει λόγος να θέσουμε κάποια ερώτηση. Ο κύριος Χουντής αλλά θα ήθελα να τελειώσουμε με τον κατάλογο και μετά σας δώσω το λόγο. Δεν θέλετε το λόγο. Ο κύριος Λούσεμπεργκ, ο κύριος Τερνέζε. Συγγνώμη, Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μιλάει με μία μόνο φωνή. Απεφάνθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει, μιλάτε με μία φωνή, αλλά υπάρχουν και διακλαδώσεις. Ο καθένας έχει και την ειδικότητά του, έχει και τις αρμοδιότητές τους και σας ζητάμε ορισμένες φορές να ε, επισέλθετε σε κάποιε λεπτομέρειε βάσει και τη εμπειρογνωμοσύνη σας. Εάν τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχουν κάποιε διαφορέ και δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πούν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων διευθύνσεων τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή να προχωρήσουμε. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ερωτήσει. Εξαιρετικά, να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Χουντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είδα τις αναφορές στις οποίες ε, τις οποίες συζητούμε, άκουσα και την επιχειρηματολογία της Κομισιόν. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε εμείς, δεν είναι θέμα της Επιτροπής Αναφορών. Απλώς θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια, τα οποία βεβαίως έχουν πολιτικό χαρακτήρα και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εμείς. Παραδείγματος χάρη, ε, προφανώς από ό,τι κατάλαβα το θέμα βρίσκεται σε επίπεδο διαιτησίας. Το κράτος της Αργεντινής ενδεχομένως επικαλείται αρχή του, βασικού, του, του, διεθνούς δικαίου η οποία λέει ότι δεν μπορώ να πληρώσω state of necessity και με βάση αυτή την αρχή λέει δεν μπορώ να πληρώσω ενδεχομένως και οι κάτοχοι των ομολόγων ζητούν τα χρήματά τους. Αυτό λοιπόν λύνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι μια γενικότερη πολιτική, η Επιτροπή Αναφορών μας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν μπορεί, ε, μάλλον Απ' την άλλη πλευρά και τελευταία μου παρατήρηση, ενδεχομένως να προετοιμαστούμε να συζητήσουμε παρόμοια περίπτωση αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι όπως θα ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρος, εκπρόσωποι της Κομισιόν, έχουμε πρόβλημα επί ελληνικού εδάφους. Με το κούρεμα των ομολόγων που έγινε με το PSI και τη Νέα Δανειακή Σύμβαση, πολλοί κάτοχοι ομολόγων του ελληνικού δημοσίου έχουν χάσει μέρος τη αξία των ομολόγων και των χρημάτων που έχουν δανείσει. Η κατάσταση είναι δραματική στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με ασφαλιστικά, ε, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Εκεί είναι σίγουρο ότι θα έρθουν διαμαρτυρίες που βρίσκονται ακόμα στο πολιτικό επίπεδο. Είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί η Επιτροπή μας θα χρειαστεί να δει κατά πόσον αυτές οι ρυθμίσεις που λαμβάνονται βεβαίως σε οικονομικό επίπεδο μέσω μνημονίων μέσω τρόικας, ας, βάλω, ας το θέσω έτσι, είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι συμβατές. Το ανέφερα απλώς σε αποστροφή ή σε αντίθεση με το ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια, με μια διένεξη με το κράτος της Αργεντινής που έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά αλλά είναι θέμα διεθνούς δικαίου και μια φωτογραφία από το μέλλον ότι πιθανό να έχουμε όχι σίγουρα τέτοιες περιπτώσεις αλλά επί ευρωπαϊκού δικαίου. Επομένως όσο αφορά τι συγκεκριμένε αναφορές νομίζω ότι η Επιτροπή μας δεν μπορεί να τις αναφέρει και πρέπει να τις ε, απορρίψει, να τις κλείσει, δεν μπορούμε να τις συζητήσουμε. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χουντή. Δεν είναι τόσο ερώτηση, αλλά θα ήθελα να σας πω κάποια σχόλια. Απευθύνομαι σε προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως να είναι χρήσιμο αυτό που θα σας πω. Προς το παρόν, από τις πληροφορίες που έχουμε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνησε ότι θα ληφθούν μέτρα κυρώσεις ε, για τις ε, σχέσεις με την Αργεντινή, ε, τα οποία μέτρα μεταξύ άλλων προβλέπουν και το κλείσιμο της έδρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αργεντινή. αυτό διότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της διαφθοράς που έχει η χώρα και αυτά είναι στοιχεία τα οποία λάβαμε από επίσημα έγγραφα και από το διεθνή τύπο φυσικά. Όλα αυτά ήρθαν φυσικά σε συνέπεια και του γεγονότος ότι δεν υπήρχε ε, διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και στις ε, δραστηριότητες που αφορούν τον προπολογισμό της χώρας. Ε, ένας μεγάλος λοιπόν διεθνής οργανισμός, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έχει φυσικά και τις ε, ιδιαίτερότητε του, αποφάσισε να αντιδράσει. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανο δεν βλέπουν πέραν της ε, λογικής ένστασης που μας εξέφρασε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το γεγονός ότι κρεμεί και μια διαδικασία διατησίας το, δεν, το οποίο δεν επιτρέπει να γίνουν άλλα διπλωματικά διαβήματα. Όπως έλεγα, δεν είναι δυνατόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όμως ε, να σιωπούν και να μην αντιδρούν καθόλου ενώπιον μιας τέτοιας κατάστασης ε, στην οποία εμπλέκονται και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Um, thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Καταγράφω τα σχόλιά σας. Θα συνεχίσουμε προφανώς να ελέγχουμε την κατάσταση για να δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις εφόσον κλείσει η διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Πρέπει να σας πω το εξής. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν δεσμεύεται από τους κανόνες διατησίας να μην επέμβει διπλωματικά. Έχει τη δυνατότητα αυτή. Και κατάλαβε επίσης ότι υπήρξε μια αντίδραση σε ένα γενικότερο συστημικό πρόβλημα το οποίο είχε εντοπίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εν λόγω χώρα. Πρόκειται λοιπόν για απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η κατάσταση βέβαια των ανθρώπων που κατέχουν τα ομόλογα είναι διαφορετική. Βάσει αντικειμενικών κριτηρίων χρησιμοποιούνται νομικά μέσα για να επιληθεί το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τους κατόχους των ομολόγων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποια θα είναι η έκβαση αυτής της νομικής διαδικασίας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόντες. Δεν θα ήθελα όμως να υπάρξει καμία σάφια στη συζήτηση. Εγώ αναφέρθηκα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν ε, έγινε όμω αυτή η αναφορά διότι ήθελα να κάνω κάποιο παραλληλισμό με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σας είπα ότι πρόκειται για κάτι εντελώ διαφορετικό. Κάθε άλλο, ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν εντελώ διαφορετικό φορέα, και η δραστηριότητα θεσμοθετές του φυσικά πόρο απέχουν από το βασικό πολιτικό ρόλο που έχουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς αναρωτιόμουν μήπως ε, επειδή ακριβώς ε, φέρθηκε έτσι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έπρεπε ίσως και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ε, δράσουν με πολιτικό τρόπο κάπως διαφορετικά από ό,τι κάνουν τώρα. Ε, όμως και το λέω εκ νέου ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει και τεχνική ένσταση που δεν επιτρέπει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ξεκινήσουν οποιοδήποτε διπλωματικό διάβιβο όταν εκκρεμεί μια διαδικασία διατησίας όπως άλλωστε προβλέπεται και στη διμερή συμφωνία μεταξύ ε, Αργεντινή και Ιταλία. Δεν ήθελα να προσθέσω τίποτα άλλο. Απλώ το είπα εν είδη διευκρίνηση. Άκουσα τι είπε ο κύριο Χουντή, ο οποίο ε, ε, επεσήμανε ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη δική μας την Επιτροπή και τι αρμοδιότητες έχει για τα σημεία αυτά και μας είπε ότι είναι περιορισμένη η δυνατότητα δράσης που έχουμε και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Νομίζω όμως ότι βάσει των δηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως θα έπρεπε να μην αφήσουμε αυτούς τους πολίτες ε, χωρίς απάντηση και να κλείσουμε σήμερα την αναφορά. Ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε, όπως είπε και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαιτησίας και από εκεί και πέρα, βάσει και το αποτέλεσμα, να αξιολογήσουμε ε, κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να παρέμβουν ε, περαιτέρω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, θα αφήσω ανοιχτά ε, τις αναφορές αυτές ε, με τη διαδικασία που σας υπέδειξα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και πάλι στους προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 11. Αναφορά 1331 του 2010, 1621 επίσης του 2010, 11-06 του 2011 και ε, 05 του 2011 και 7-99 του 2011. Τις εξετάζουμε όλες μαζί διότι ε, είναι κοινό το αντικείμενό τους. Σήμερα ε, υπάρχουμε ε, κάποιοι εκ των αναφερόντων. Ο κύριος Μάριο Ντεκρεσέντσο, εκπρόσωπος ε, της ε, ε, Ένωσης Μομπάστα, φτάνει πια, στον οποίο φυσικά θα δώσω και το λόγο για να μας εξηγήσει λίγο το ζήτημα. Να υπενθυμίσω βέβαια όμως ότι έχει γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής αφιερωμένη στο ζήτημα και ελπίζω να έχουν εξελιχθεί λίγο τα πράγματα. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε πέρασαν ακριβώς 18 χρόνια στην ε, Ιταλία από τότε που ετέθησε ε, εφαρμογή οδηγία 9249 και θεωρώ ότι θα πρέπει να σας δώσω μια εικόνα για τις τιμές ε, ασφαλιών αυτοκινήτων στην Ιταλία. Στην Ιταλία πληρώνουμε τιμές ρεκόρ για την ασφάλεια των αυτοκινήτων μας, σχεδόν διπλάσιες από το κόστος των ασφαλιστικών συμβάσεων στη Γερμανία, στην Ισπανία και στη Γαλλία. Ε, για, κατά μέσο όρο πληρώνεται ε, ασφάλιστρα ε, 400 ευρώ, στη Γερμανία 222, στη Γαλλία 172 και στην Ισπανία 229 ευρώ. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι ανησυχητική η κατάσταση και επιβεβαιώνει ότι η Ιταλία δεν προσαρμόστηκε στην πράξη στην ε, οδηγία αυτή. Αλλά στην Νότια Ιταλία αυτή η διαφορά γίνεται παράλογη τελείως, διότι εκεί οι τιμές είναι τρεις ή τέσσερις φορές υψηλότερες από τις υψηλότερες τιμές που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ιταλία. Πρόκειται ουσιαστικά λοιπόν για κόλαφο κατά της ε, απελευθέρωσης και της διαφάνειας που προτίθεται το 1994. Ε, ο πρώτο πραγματικός παραλογισμός προκύπτει αμέσω. Η μεγάλη διαφορά των τιμών από κάθε, σε κάθε περιφέρεια θα έπρεπε ε, να δοθεί με στατιστικά στοιχεία και να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για τους καταναλωτέ. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται στην Ιταλία. Καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα κανένα στατιστικό στοιχείο, ούτε σε εθνικό αλλά ούτε και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μια στάση την οποία θα πρέπει να τιμωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από τότε που ξεκίνησε η κοινή αγορά ε, ήμασταν πάντα υπέρ τη διαφάνεια προ όφελο του καταναλωτή. Κάτι το οποίο έχουν λησμονήσει πλήρω οι ασφαλιστικέ εταιρείε στην Ιταλία. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η θέση της ε, Άνια, της ε, ε, Εθνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Η ένωση αυτή ισχυρίζεται ότι ε, υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά ε, στις ε, νότιες περιοχές της Ιταλίας. Όπως σας είπα όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στατιστικό στοιχείο, γεγονός που επηρεάζει την αγορά των ασφαλιών ε, στην Ιταλία, διότι δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που να βγαίνει από αυτό το καρτέλ το οποίο είναι προφανές. Η δήλωση στη Σάνια είναι ε, σε σαφή αντίθεση με τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε, τα στοιχεία του ISVP και τα έχουμε αποστείλει εδώ στην Επιτροπή σας. Και προκύπτει ένα σενάριο το οποίο είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ε, δεν υπάρχουν διαφορές ε, στις τιμές μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ιταλίας, κυρίως μεταξύ Βορρά και Νότου. Ε, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ε, την περιοχή της Νάπολη, θα δείτε πόσο διαφορετικά άλλαξαν τα πράγματα από το 2009 στο 2010 και λέει ότι οι τιμές στην Νάπολη είναι χαμηλότερες από το Μιλάνο, αλλά παρόλα αυτά στην Νάπολη οι εταιρείε εφαρμόζουν ε, τιμές 30% περισσότερο από ό,τι στο Μιλάνο. Ε, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία. Δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια στις πληροφορίες που λαμβάνουμε και κυρίως επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει πραγματικό καρτέλ το οποίο ε, γίνεται πλέον ρατσισμός ασφαλιστικής φύσεως. Και αυτό προκύπτει από τα όσα συνέβησαν από μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Δήμο της Νάπολης που λέγεται «Έρεση Άουτο Νάπολη Βουρτουάζα». Ε, προσπαθώντας να επιτύχουμε χαμηλότερες τιμές, η ασφαλιστική εταιρεία πρότεινε ε, μία μετατροπή που απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία. Ο Δήμος απάντησε ότι οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να ασφαλιστούν θα πρέπει να μην έχουν ε, δημιουργήσει ατυχήματα, να έχουν πληρώσει τις φόρους τους ε, και να μην υπάρχει πρόβλημα κανένα με το κράτος. Ουσιαστικά να είναι ε, πρότυπο ε, πολιτών. Και όμως μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων μόνο μία ασφαλιστική εταιρεία μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, η Admiral που είναι αγγλικών συμφερόντων και ούτως ή άλλως οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές σε σχέση με το μέσο όρο που έχουμε σε εθνικό επίπεδο. Το θέμα είναι ότι ε, ασκώντας πιέσεις προς την πολιτική, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καταφέρουν τελικώς να καθορίσουν αποφάσεις οι οποίες είναι ε, βάση ε, των απαιτήσεων των ισχυρών και όχι υπέρ των πολιτών. Το πιο κατάφορο παράδειγμα της ε, ε, επιρροής που έχουν ασφαλιστικές εταιρείες στην Ιταλική πολιτική είναι αυτό το οποίο συνέβη μετά από την θέση σε ισχύ της λεγόμενης απόφασης της απελευθέρωσης, το οποίο έγινε νόμος στα τέλη Μαρτίου και εκεί ε, προτάθηκε ουσιαστικά ε, στις ε, ασφαλιστικές εταιρείες μια σειρά από κανόνες που θέλουν να μειώσουν την απάτη. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει αποζημίωση για ζημία η οποία προκαλείται από πρόσκρουση και υπάρχουν και κάποιες ποινές οι οποίες καταργούνται όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις για ασφαλιστικές απάτες. Ουσιαστικά ε, προσπαθούν να βάλουν στα αυτοκίνητα ένα μαύρο κουτί το οποίο θα επιτρέπει ε, να μην υπάρχουν ε, προβλήματα και την εφαρμογή του άρθρου 32 που λέει, και σας παραθέτω, ότι για τις κατηγορίες τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση, βάσει υποκειμενικών και αντικειμενικών συνθήκων, η κάθε μία από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να προτείνει αντίστοιχες προσφορές. Ε, αν δούμε και όλα όμως ε, τα ωφέλη της ε, ε, νομοθεσίας κατά της απάτης, όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είπαν ότι δεν θέλουν να εφαρμόσουν κανένα από τα μέτρα τα οποία είναι προς όφελος των καταναλωτών. Μετά από τρεις μήνες κανένα από αυτά τα σημεία δεν έχει εφαρμοστεί. Όσον αφορά την έκπτωση που αφορά τα ασφάλιστρα, ε, λέει ότι αυτά καταργούνται από την αύξηση που θα υπάρξει με την ε, εκπνοή της ε, ασφαλιστικής υπηρεσίας. Όσον αφορά αυτό το μαύρο κουτί, δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα πρέπει να εφαρμοστούν και επομένως πώς θα υπάρχει η έκπτωση εάν δεχτούν οι αυτοκινητιστές να έχουν αυτό το μαύρο κουτί στο αυτοκίνητό τους. Αλλά το βασικό σημείο του σημείο 3, το οποίο δίνει μεγάλη ισχύ στις ασφαλιστικές εταιρείες και το, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ε, διαφορές στις τιμές μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ιταλία, αλλά παρόλα αυτά ε, δηλώνει ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστούν οι κοινοτικοί κανόνες, λέγοντας ότι το άρθρο 6 της Οδηγίας 9249 είναι ανεφάρμοστο. Το άρθρο 6 λέει ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν καθορίζουν διατάξεις που αφορούν την προηγούμενη έγκριση των γενικών και ειδικών συνθηκών των ασφαλιστικών εταιριών. Ουσιαστικά δεν πρέπει να γίνει η πρώτερη έγκριση των τιμών και επομένω η κάθε ασφαλιστική εταιρεία, η κάθε μία δηλαδή, μπορεί να εφαρμόσει σεβόμενη και φυσικά τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, την τιμή που θεωρεί πιο δίκαιη η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία και ξεχνούν την αρχή της ισότητας βάσει της οποίας δύο πολίτες που είναι οι ίδιοι οδηγοί, αλλά ζουν σε διαφορετικές ε, πόλεις, ε, πρέπει να πληρώνουν το ίδιο τίμημο, το οποίο ε, σφέρει και η Ιταλική νομοθεσία. Στο σημείο 8 τώρα, στην ίδια κινητική νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα κάθε κράτο μέλο να εφαρμόζει πιο περιοριστικού κανόνε για τι ασφαλιστικέ εταιρείε. Γεγονό το οποίο θεωρούμε ότι συνάδει με το ε, σημείο 3,2 ε, ε, του διατάγματος που υπήρχε για την ε, απελευθέρωση των αγορών που σας είπα. Επίσης θεωρούμε ότι δεν έχει επιτύχει η μεταφορά της οδηγίας στην Ιταλική νομοθεσία και η ε, ε, αυτοκινητοβιομηχανίες ε, είναι πλέον ε, σχεδόν στα πρόθυρα της καταστροφής. Πολλές έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν και χάνονται λοιπόν και θέσεις εργασίας και σε συνεργεία και σε αυτοκινητοβιομηχανίες. Επομένως εγκαταλείπεται σχεδόν ε, ε, η περιοχή και χάνονται και εκεί θέσεις εργασίας. Είναι αδύνατον από πλευράς νέων να οργανώσουν εργατικές δραστηριότητες που προβλέπουν χρήση αυτοκινήτων, διότι ένας νέος οδηγός ε, στην Νότια Ιταλία πρέπει να πληρώνει 4.000 ευρώ το χρόνο για ασφάλιστρα για το αυτοκίνητό του. Αυτά όλα είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση για όλες τις Ιταλικές ε, οικογένειες ε, στο νότο της Ιταλίας και πολλές φορές αναγκάζονται να πουλήσουν το αυτοκίνητό τους διότι δεν μπορούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτό φυσικά ε, είναι εις βάρος του συλλογικού κοινού καλού. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νάβα, τον Διευθυντή, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ και ελπίζω να μπορέσει να μας βοηθήσει για να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία θέσαμε στον Επίτροπο Μπαρνιέ για το θέμα αυτό το οποίο μόλις μας παρουσίασε ο αναφέρον. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εν συντομία ποια είναι η ερώτηση. Ζητάμε καταρχάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κατά πόσο λυθεύει η έκκληση που έκανε ο Ιταλός υπουργό ε, σε απάντηση στα θέματα τα οποία ε, τέθησαν και στην Ιταλική κυβέρνηση ότι η στάση λοιπόν της Ιταλικής κυβέρνησης όπως το κατήγγυλαν οι αναφέροντες και επιβεβαιώθηκε και από τον ε, Ιταλό νομοθέτη σε πρόσφατη παρέμβασή του οφείλεται σε ε, λανθασμένη ερμηνεία της 92 ε, 49. έχουμε επισυνάψει την απάντηση του Υπουργού και της ε, Άνια και της ε, ISVAP που χρησιμοποίησαν αυτή την αναφορά για να απαντήσουν αρνητικά στις καταγγελίες που έχουν κάνει οι Ιταλοί πολίτες και που ακούσαμε σήμερα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Διευθυντή, τον κύριο Νάβα, τον οποίο ευχαριστώ εκ νέου για την παρουσία του. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κυρία Ματσόνη. Καλημερίζω και τους αναφέροντες. Θα μιλήσω Ιταλικά, διότι είναι προς όφελος και των ε, ε, επιτρέψτε μου, διότι υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία έθιξαν οι αναφέροντες και είναι πολύ ενδιαφέροντα και ίσως θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε λίγο και τη συζήτηση για το θέμα αυτό. δεν να σας πω ότι συμφωνώ κυρίως με τα τελευταία σημεία τα οποία μας θίξατε, δηλαδή τι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την κατάσταση. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω μαζί σας είναι να προσπαθήσουμε να βρίσκουμε ποια είναι η ουσία του προβλήματος, ποια μπορεί να είναι τα αίτια, αλλά σίγουρα συμπάσχω με τα όσα ακούστηκαν ε, στο τέλος ε, και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο θέσεων απασχόληση. Ε, πρώτο και κυριότερο, άρθρο 6 τη οδηγία. Υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ε, επιβεβαιωμένη νομολογία. Η 346 του 2002 και η 347 του 2002 και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λέει σαφέστατα ότι βάσει στοιχείων οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να θεωρήσουν διαφορετικούς ε, ε, παράγοντες κινδύνου και μπορούν να καθορίσουν και ότι ο τόπος διαμονής είναι στοιχείο διαφοροποίησης. Ε, μπορεί να υπάρχει λοιπόν κίνδυνος λόγω του τόπου διαμονής κάποιου. Αυτό βέβαια είναι μόνο μερικός η απάντηση. Από νομική σκοπιά λοιπόν είναι ορθό να πούμε ότι μπορεί κάποιος να επιβάλλει ε, μια συγκεκριμένη τιμή στα ασφάλιστρα... Ε, με ένα παράγοντα κινδύνου τον οποίο αντικειμενικά αναγνωρίζουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα τον τύπο του αυτοκινήτου. Ε, ανάλογα με τον ε, ε, τύπο του αυτοκινήτου είναι διαφορετικός ο παράγοντας κινδύνου, ε, το παρελθόν φυσικά του ασφαλισμένου και ούτω καθεξής. Ε, μαζί όμως με αυτό υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία κατεμέτα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η νομική διάταξη, όπως σας είπα, είναι διότι πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων κινδύνου που επιτρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη προσφορά διαφόρων ε, ασφαλιστικών συμβουλέων. Αυτό το οποίο όμως μας ε, έθιξαν οι αναφέροντες είναι νομίζω πέραν αυτής της πτυχής. Διότι ναι μεν υπάρχει το θέμα της διαφοροποίησης, αλλά αφετέρου υπάρχει και ως προς τι ε, κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας το απέδειξαν οι αναφέροντες και επίσης αυτή τη στιγμή έχει καθοριστεί προς ως γίνεται η διαφοροποίηση, ποιο είναι το ποσό το οποίο αιτιολογεί αυτή τη διαφοροποίηση. Αυτές, κατά την άποψή μου, είναι δύο πτυχέ τις οποίες θα πρέπει να επισημάνουμε. Οι αναφέροντες λένε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία από πλευράς ασφαλιστικών εταιριών και είναι σαφές ότι, ότι η κάθε ασφαλιστική εταιρεία θεωρεί ότι το χαρτοφυλάκιο των πελατών της ε, και τα στοιχεία τα οποία θεωρεί παράγοντες κινδύνου είναι ε, ιδιωτικά στοιχεία και αφορούν την εμπειρογνωμοσύνη τη, αλλά σε σεβαίωμενοι και αυτό το ιδιωτικό στοιχείο και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν και εμπορικά μυστικά, υπάρχει τρόπος ε, να... έχουμε στατιστικά στοιχεία, διότι επειδή μιλάμε για τον τόπο διαμονής, θα μπορούσε ίσως να εξευρεθεί ένας μηχανισμός να μπορούμε να κρατήσουμε απόρριτα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την κάθε ασφαλιστική εταιρεία, αλλά να δείξουμε ποιο είναι το στοιχείο του κινδύνου το οποίο προκύπτει λόγω ε, ενός συγκεκριμένου γεωγραφικού σημείου, ενός, του τόπου διαμονής κάποιου. Είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε και θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία μπορούν να μας επιτρέξουμε να αξιολογήσουμε ε, αντικειμενικά τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του τόπου διαμονής των ασφαλισμένων. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά ε, και να υπάρχουν κάποια απόρριτα στοιχεία, αλλά υπάρχει και μια αντικειμενική διαφορά την οποία μπορούμε να ε, εξετάσουμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ενστάσεις ε, σε μεμονωμένο επίπεδο, αλλά σε επίπεδο συνόλου, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία. Και αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν είτε οι αρχές, είτε ε, μια πρωτοβουλία πολιτών, όπως η άλλη πρωτοβουλία που αναφέρθηκε. Ε, μια δεύτερη πτυχή, την οποία μας ανέφεραν οι αναφέροντες, είναι ότι έστω ότι λαμπτυχία, στοιχεία, ποιο ποσό διαφοροποίησης δικαιολογείται βάσει στατιστικών στοιχείων. Και εδώ νομίζω ότι ε, επίσης ε, υπάρχουν πολλά να γίνουν, διότι Κανεί δεν μπορεί να καταχράτε μια πιθανή διαφοροποίηση. Άλλο είναι να λέμε ότι γίνεται διαφοροποίηση και άλλο να γίνεται κατάχρηση λόγω αυτής της διαφοροποίηση. και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο ανέφεραν ε, οι αναφέροντες είναι οι τελευταίοι κανόνες, οι τελευταίοι νόμοι που εισήχθησαν. Νομίζω ότι και εδώ στην αίθουσα αλλά και εκτός αιθούση, συμφωνούμε όλοι ότι όταν ε, εισάγονται νόμοι οι οποίοι στόχο έχουν τη μείωση της απάτης, ε, σίγουρα είναι πρόσδεκτοι. Είναι σίγουρα λοιπόν ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι υπάρχουν μια σειρά από κανόνες ε, που αυξάνουν τις ε, ε, κυρώσεις που ζητούν να υπάρξει αυτό το μαύρο κουτί και ούτω καθεξής. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό οι αρχές και σε αυτή την περίπτωση να εξετάσουν πάρα πολύ καλά πώς θα γίνει το πέρασμα και είχε προβλεφθεί μια δοκιμή, ένα στόχος. Ο στόχος είναι η μείωση της απάτης. Είναι η ε, δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερη αποπτή από πλευράς ασφαλιστικών εταιριών και μέσω αυτού να μειωθούν ίσως και τα ε, ασφάλιστρα. Αυτά λοιπόν κατ' είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως βάση εργασίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Οδηγία 9249 ήταν εν γέννη ε, ωφέλιμη. Το γεγονός ότι περάσαμε σε απελευθέρωση τιμών και δεν είχαμε ε, ρύθμιση των τιμών σίγουρα είναι κάτι το ωφέλιμο. Αλλά εάν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι διαφορές δεν βασίζονται ούτε σε αυτά στοιχεία, ούτε αιτιολογούνται με κανένα τρόπο και αυτές οι περιπτώσεις είναι ε, μεταξύ διαφόρων νομών ή επαρχιών ή περιφερειών όπως λένε οι αναφέροντες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ριβελίνη. Πολύ σύντομα, ευχαριστώ την Επιτροπή, τον κύριο Νάβα. Αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συζητάμε. Και θα ήθελα σεβόμενοι και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, να διευκρινίσω το ζήτημα. Κύριε Νάβα, εδώ έχουμε ρατσισμό ε, εις βάρος των πολιτών του Νότου της Ιταλίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν εγώ διαπράξω ένα αδίκημα και το ίδιο αδίκημα το κάνει και ο κύριος Βαλέσα στην Πολωνία, ο δικαστής πρέπει να με καταδικάσει, όχι γιατί μένω σε ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά για το έγκλημα ή το αδίκημα που διέπρεξα. Και σας ρωτώ, και εδώ θα ήθελα μια σαφή απάντηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο πολίτες νέοι οδηγοί, που μόλις πήραν το δίπλωμά του και δεν έχουν ακόμα ε, ποινικό μητρό εντό εισαγωγικών στην οδήγηση, διότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει την εντύπωση στην ασφαλιστική εταιρεία ότι είναι κακή οδηγή. Δύο νέοι οδηγοί. Ένας που γεννήθηκε στην Νάπολη και μένει στην Νάπολη και ένας που μένει στο Μιλάνο. Έχουν μια διαφορά σε ασφάλιστρα και αυτός που μένει στην Νάπολη πληρώνει το εξαπλάσιο ή το επταπλάσιο. Δύο πολίτε που δεν έχουν τίποτα. Είναι κενό το διπλωμά του, δεν υπάρχει κανένα πτέσμα διότι μόλι το πήρανε. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν προασπίσει τα δικαιώματά του, ε, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κινέζων, των Αφρικανών και δεν προασπιζόμαστε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, διότι αυτά είναι δικαιώματα. Δύο πολίτε που μόλις πήραν το δίπλωμά τους, που δεν έχουν οδηγήσει πουθενά, έχουν δύο διαφορετικές τιμές ασφαλίστρων, απλώς και μόνο γιατί μένουν σε άλλη πόλη. Αν αυτό δεν είναι διάκριση, πέστε μου εσείς πώς τη λέμε. Και εγώ ως Ευρωπαίος πολίτης, όχι πολίτης του Νότου της Ιταλίας, έχω σκοπό να προχωρήσω στη μάχη αυτή μέχρι τέλους. Και πραγματικά ελπίζω όλοι οι βουλευτές, από όλες τις χώρες, από όλες τις πολιτικές ομάδες, να υπερασπιστούν αυτό το όνειδος και να παρέμβουν το συντομότερο δυνατόν. Διότι πρέπει να πάψει να υπάρχει αυτός ο ρατσισμός και πρόκειται για ρατσισμό ενώπιον των ε, νοτίων Ιταλών. Ε, Σα ευχαριστούμε κύριε Ριβελίνη. δεν υπάρχει κανεί άλλος που θέλει το λόγο, κύριο Νάου. Ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω Άλλο είναι το έγκλημα. Αν οι δύο νέοι οδηγοί που είπατε εσεί ε, πατήσουν και οι δύο με το αυτοκίνητό του κάποιον, σίγουρα και οι δύο διαπράττουν ένα δίκημα και πρέπει να τιμωρηθούν αναλόγω. Άλλο αυτό και άλλο ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι δύο νέοι οδηγοί ο τύπος του κινδύνου δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός ότι βρίσκονται υπό ίδιες προϋποθέσεις αυτοί οι δύο νέοι οδηγοί, αλλά αφορούν και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται αυτοί οι δύο ε, νέοι οδηγοί. Αν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνο σε μια περιοχή σε σχέση με μια άλλη, δεν είναι παράλογο να υπάρχει διαφορά μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών. Αυτό το οποίο είναι παράλογο και επ' αυτού επιμένω, διότι εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι ότι αυτοί η διαφορά του κινδύνου δεν αποδεικνύεται ούτε ότι υπάρχει, αλλά ούτε στο ποσό της διαφοροποίησης. Δεν είναι αιτιολογισμένο αυτό το ποσό. Διότι αν είναι διπλός ο κίνδυνος, για παράδειγμα, ε, τυχαίο παράδειγμα σας δίνω, αν είναι λοιπόν διπλός ο κίνδυνος, τότε ε, θα μπορούσε να είναι διπλό το τίμημα των ασφαλίστρων. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε. Αλλά ε, δεν θεωρείται παράλογο να θεωρούνται διαφορετικά τα επίπεδα κινδύνου σε κάθε περιοχή και να υπάρχει και διαφορετικός κίνδυνος. Αυτό είναι κάτι το οποίο ζούμε όλοι μας, ε, στον καθημερινότητα εξαρτάται και από τον κίνδυνο. Αν κάποιος είναι καπνιστής πληρώνει περισσότερα, αν δεν είναι καπνιστής πληρώνει λιγότερα. Υπάρχει λοιπόν και ένα ευρύτερο περιβάλλον το οποίο πρέπει να βάλουμε υπόψη. Αλλά το ποσοστό της διαφοροποίησης είναι αυτό στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ε, για να απαντήσουν οι αναφέροντες. Κύριε Νάβα, καλημέρα. Το πρόβλημα το οποίο θίξατε αφορά τα σύνολα των δεδομένων τα οποία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ε, ότι αν κάνουμε σύγκριση κάποιες αστικές περιοχές, για παράδειγμα την περιοχή της Νάπολης και του Μιλάνου, έχουμε ενδείξεις ότι τα επίσημα στοιχεία αναφέρονται σε διαφορά κόστους μεταξύ των ασφαλίστρων και του κινδύνου κατά 2,30% επιπλέον. Δεν εξηγείται λοιπόν όλα όσα συμβαίνουν αργότερα. Παραδείγματο χάρη, να υπάρχει μια διαφορά στη τιμή κατά 50 περίπου 100. Αυτό επαληθεύεται με τους ελέγχους του οποίους αναφέρετε κι εσείς, οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν. Και ολοκληρώνοντας, το μόνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ο Ιταλικός νόμος δεν έδωσε τη δυνατότητα στον Επιπτικό φορέα να επαληθεύσει επακριβώς με ποιο τρόπο εφαρμόζονται οι διάφοροι νόμοι. Ολοκληρώνω ένα τελευταίο στοιχείο. Στην Ιταλία οι ασφαλιστικές εταιρείε μπορούν να ακυρώσουν τα ασφαλιστικά συμβόλαια με τους ε, ε, πολίτες μέσα σε 30 ημέρες. Οι πολίτες μπορούν να απαντήσουν ε, εντός 45 ημερών. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο ίδιος ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα ε, στον πολίτη να δώσει κατάλληλη απάντηση ώστε να διορθώσει μια κατάσταση η οποία έχει προκύψει από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέσει μια ασφαλιστική επιχείρηση για να ασφαλίσει έναν πολίτη του Νότου της Ιταλίας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Διευθυντής ε, του Επιτρόπου Μπαρνέ μας έδωσε μια καλή άγουσα πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Εγώ ε, θα... Ε, ακούσω και στο διαδίκτυο τις παρεμβάσεις σας για να έχω λέξη προς λέξη τα όσα είπατε. Είδαμε και πώς συμπεριφέρεται η εθνική νομοθεσία και αν δικαιολογούνται αυτές οι διαφορές μεταξύ των χωρών. Η οδηγία βέβαια στην οποία αναφέρθηκε ο Υπουργό επιτρέπει τι διαφορέ, αλλά όπω μα είπε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τι δικαιολογεί. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο σημείο αυτό όταν θα έχουμε εξετάσει ακριβώ τι μα είπε ο ε, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν ενστάσει από πλευρά συναδέλφων, θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά διότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε το ζήτημα βάσει των παρατηρήσεων και που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχουν ενστάσεις, επομένως ε, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα αυτό και ευχαριστούμε και τους αναφέροντες. Περνάμε τώρα στο σημείο 12. Έχουμε δύο αναφορές εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών. Για το σημείο αυτό ε, έχουμε κάνει συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή μας. Έχουμε φτάσει μέχρι και στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, όπου είχαμε την έγκριση ενός ψηφίσματος πολύ σημαντικού για τη σύναψη της Διεθνούς ε, Συμφωνίας ε, για τη δημοσίευση ε, βιβλίων σε μπράι για να μπορούν να τα διαβάσουν τα τυφλά άτομα και σήμερα έχουμε ζητήσει να ε, παραστεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να μας ενημερώσει για το ε, τι ακριβώς συνέβη μετά από τη συζήτηση στην οποία αναφέρθηκα. Να δώσω λοιπόν απευθεία το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου για να μας ε, ενημερώσει και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε και τους συναδέλφους. Good morning everybody. I am... Είμαστε ευγνώμονες και σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας σήμερα να παραστούμε. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για εκείνους που τους στερείται αυτό το δικαίωμα που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους να μπορέσουν να έχουν στη διάθεσή τους αυτό που όλοι έχουμε ως ικανότητα Είμαι όμως βέβαια ότι έχουν άλλα δώρα και προσόντα που δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι οι κανονικοί άνθρωποι. Του του η Κυπριακή Προεδρία πραγματικά δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Επίσης είναι σημαντικό ζήτημα για μας. Και προτού καν αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου, με την Δανέζικη Δανική Προεδρία στο παρελθόν είχαμε παρακολουθήσει όταν μας προσκάλεσε στη Γενέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άτυπες συζητήσεις για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του μηνός Μαΐου. Είχαμε συμμετάσχει έτσι. Και μετά, συγγνώμη, λίγη ησυχία παρακαλώ, τι γίνεται εδώ. Μιλάνε εκεί πίσω, δεν μπορώ πραγματικά να συνεχίσω. Συγγνώμη, δεν μπορώ λέω να συνεχίσω έτσι και δεν μπορώ να εκφραστώ με αξιοπρεπή τρόπο μέσα σε αυτό το χάος. Λοιπόν. Okay, sorry for this. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ λοιπόν και ζητώ συγγνώμη. Αλλά είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις ηχητικές και δεν μπορούσα να συνεχίσω και να συγκεντρωθώ. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτό που προσπαθούσα να πω πιο πριν είναι ότι πραγματικά είμαι ευγνώμων για την πρόσκλησή σας και με ιδιαίτερη προσοχή στρέφουμε τα μάτια μας σε αυτό, την προσοχή μας σε αυτό το θέμα και ως Κυπριακή Προεδρία. Παρίσταμε σήμερα για να ακούσω, να αφουγκραστώ τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας που θα θέλατε να κάνετε προς εμάς την Κυπριακή Προεδρία και να σημειώσω όλες τις προτάσεις και σχόλιά σας. Αν έχετε ήδη ή αν είσαστε παρόντες ή παρούσες στην νομική επιτροπή προ, ε, προχθές, ο Προεδρεύων, ε, πρόεδρος του Συμβουλίου χθες όταν παρουσίαζε, προχθές όταν παρουσίαζε τις, προ, τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας ρητά και κατηγορηματικά αναφέρθηκε στο θέμα αυτού του σχεδίου συνθήκης ε, ή σχεδίου μέσου που ε, βρίσκεται υπό συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει ήδη εξετάσαμε αυτό το έγγραφο, τον τίτλο σε σχέση με τα κράτη-μέλη και την εμπλοκή τους για την δημιουργία ενός διεθνούς μέσου για άτομα που έχουν προβλήματα όρασης. Ήδη κατά την πρώτη ομάδα εργασίας που είχαμε συνέρθει σε αυτήν στις 5 του μήνα Ιουλίου. Ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις σε αυτή τη φάση και έχουμε υπόψη να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα για την επόμενη συνάντηση ε, της ομάδας εργασίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την πρόσκλησή σας. Τίνω ευήκο αότα, ευήκο νους και ευήκο αότα για να παρακολουθήσω τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ εσάς για την παρέμβασή σας και στη συνέχεια θα αρχίσουμε με τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Πρώτα, απ' όλα στους συντάκτες ε, των, της αναφοράς. Έχετε πέντε λεπτά περίπου για τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, που μας δώσατε την δυνατότητα να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Θέλω να παρατηρήσω ότι τρεις οργανώσεις είναι εδώ που εμπλέκονται και είναι παρούσες σε αυτό το θέμα η Ένωση Δυσλεκτικών και έχουμε τον Αντιπρόεδρο εδώ ε, και τον Chris ε, Friend από την ε, Ένωση Τυφλών και εγώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών σε σχέση με αυτή την αναφορά. Χωρίς να χρονοβορήσουμε, επειδή πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο Chris Friend, που είναι πρόσωπό και, και επικεφαλής σε αυτή την εκστρατεία εξ ονόματός μας. Κυρία Πρόεδρε, ε, μέλη της Επιτροπής Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ένωση Τυφλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμά θερμότατα την πρόσκλησή σας ε, να επανέλθουμε ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε σε σχέση με τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί και από πλευρά Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από τότε που καταθέσαμε τον Οκτώβριο πέρυσι στην Επιτροπή σας αυτή την αναφορά μας. Όπως είπε ο φίλος μου πιο πριν, έχουμε ως συν, συντάκτη την ε, Ένωση Δυσλεκτικών και εγώ εξ ονόματος και των δύο ενώσεων μας θα λάβω τον λόγο τον Φεβρουάριο ο Επίτροπος ε, για την Εσωτερική Αγορά Μισελ Μπαρνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντώντας σε μια προφορική ερώτηση από αυτήν την, σε σχέση με αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή υποσχέθηκε ότι θα ζητούσε εντολή από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπραγματευτεί μια δεσμευτικού χαρακτήρα συνθήκη για τους ε, ε, με προβλήματα όραση και ε, για τους ανθρώπους με αυτά τα προβλήματα. Υποσχέθηκε ότι θα είχε διάλογο με κάθε κράτος μέλος για αυτό το θέμα προλιένοντας ε, το έδαφος για το επίσημο αίτημα σε σχέση με το Συμβούλιο για μια διαπραγματευτική εντολή, για μια δεσμευτικού χαρακτήρα συνθήκη. Σήμερα προσβλέπουμε ακριβώς το να ακούσουμε ποια πρόοδο έχει σημειώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο Επίτροπος σε σχέση με αυτές τις δύο δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Θα θέλαμε επίσης ιδιαίτερα να ακούσουμε την ακριβή διατύπωση από πλευράς κειμένου που συμφωνήθηκε για αυτή την διαπραγματευτική εντολή ώστε να ανταποκριθούν οι υποσχέσεις ε, που έδωσε ο Επίτροπος στο Ευρωκοινοβούλιο να υλοποιηθούν σαφώς τα ίδια τα αιτήματα και οι επιθυμίες του ίδιου του Ευρωκοινοβουλίου και να ανταποκριθούν έτσι και να ε, δώσουν ε, σάρκα και οστά στις επιθυμίες εκατομμυρίων πολιτών. Αυτό πρέπει να κάνει λόγο λοιπόν ως εντολή, αυτή η εντολή πρέπει να κάνει λόγο για μια δεσμευτική συνθήκη Πρόεδρε, όταν είχα την τιμή τον προηγούμενο Οκτώβριο πέρσι να προσφωνήσω τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, κοινοποίησα, σας παρουσίασα ένα όραμα, ότι δηλαδή στις ε, δικές σας εκλογικές περιφέρειες ε, πηγαίνοντας ε, στις λεωφόρους για να μπείτε σε ένα βιβλιοπωλείο και όταν θα συναντούσατε για παράδειγμα 95% απροσδόκητα όλων των βιβλίων που δεν θα μπορούσατε να τα πάρετε να τα διαβάσετε. Από τους, στους εννέα μήνες από τότε που είχαμε την παρουσίαση της αναφοράς μας τον Οκτώβριο, πάνω από 750.000, 750.000 νέα βιβλία τυπώθηκαν, καινούργια βιβλία. Όμως μόνο 3.750 από αυτά θα είναι ποτέ στη διάθεση των τυφλών και θα είναι στη διάθεσή τους ε, στο αλφάβητο Braille για να μπορούν εκείνοι να τα διαβάσουν και να τα απολαύσουν. Σας υπενθυμίζω αυτό το σημείο πρόεδρε επειδή την επόμενη εβδομάδα στα θέματα της εξέτασης της Επιτροπής για πνευματικά, ε, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και copyright θα επομιστείτε από κοινού με τα κράτη-μέλη, με άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το προγραμματισμένο σχέδιο για την Επιτροπή για το copyright, για τα πνευματικά δικαιώματα, να ολοκληρώσετε τελικά αυτό το νομικό κείμενο και να συμφωνήσετε για τη φύση και μορφή του μέσου που θα λάβει αυτό το ε, εργαλείο για να αρχίσει να ισχύει. Τώρα, για το έργο και την επικοδομητική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πώς θα γίνει εφικτό σε αυτή τη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσετε, να κάνετε να υποβάλλετε μια σύσταση στη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου, να συγκληθεί μια διπλωματική συνδιάσκεψη το 2013. Αυτή η διπλωματική διάσκεψη θα ολοκληρώσει μέσα σε ένα σαφές πλαίσιο μια νομικά δεσμευτικά συνθήκη για τους ε, έχοντες προβλήματα όραση και εκείνους που δεν μπορούν να διαβάσουν βιβλία, τυπωμένα βιβλία. Αν αποτύχει αυτή η συνδιάσκεψη, ένας ακόμα χρόνος θα περάσει και θα χαθεί άλλα ένα εκατομμύριο βιβλία θα έχουν τυπωθεί χωρίς να έχουμε εμείς πρόσβαση σε αυτά. Γιατί δεν θα υπάρχει νόμος ή νομοθεσία που να μας επιτρέψει να αντιστρέψουμε αυτή την, αυτό τον λοιμό ε, βιβλίων που ισχύει ως κατάσταση εις βάρος μας. Εμείς ε, αυτά τα μέλη αυτής της κοινότητας που έχουμε προβλήματα όρασης ε, πραγματικά δημονούμε να επιληθεί το θέμα αυτό. Έχει εγγραφεί αυτό το θέμα από το 1982 σε σχέση με την ημερήσια διάταξη εργασιών της UNESCO και του ΟΗΕ είχαμε αυτή την προσέγγιση και τις συστάσεις από τη UNESCO να υπάρχει ένας διεθνώς δεσμευτικός νόμος για την παραγωγή και την συνολική παγκόσμια διανομή σε ειδικού, ειδικών διαστάσεων βιβλία για τους ε, έχοντες πρόβλημα όρασης. Από τα μέσα του 1980 η κοινότητα των εχόντων προβλήματα όρασης αυξήθηκε σημαντικά και συνεχίζει να αυξάνεται κάθε μέρα ο αριθμός των μελών μας, καθημερινά. Σήμερα υπολογίζουμε ότι έχουμε 438 εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά με προβλήματα όρασης με περιορισμένη όραση που εξαρτώνται από την έγκραση, έγκριση αυτής της συνθήκης για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Κυρία Πρόεδρε, εσείς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής και πράγματι όλοι οι Ευρωβουλευτές ε, έχετε αναγνώστες που έχουν προβλήματα όρασης στις δικές σας εκλογικές περιφέρειες. Κάθε φορά που φεύγετε από τις Βρυξέλλες και επιστρέφετε στις εκλογικές σας περιφέρειες, ο δικός τους αριθμός έχει εντωμεταξύ αυξηθεί. Γίνονται περισσότεροι καθημερινά συμπερασματικά. Εσείς έχετε ε, ρόλο πραγματικά θεμελιώδη που μπορείτε να διαπραγματεύσετε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Σχέδια κειμένων έχουν ε, εξεταστεί και προταθεί εδώ και τρία χρόνια πια. Τώρα πρέπει να αναλυφθεί η δράση επιτέλους. Την επόμενη εβδομάδα η Ευρώπη θα έχει μια αυθεντική πραγματική ευκαιρία να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει την επιρροή της ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η συνθήκη για τους έχοντες προβλήματα όρασης. Η Ένωση Τυφλών και οι δυσλεξικοί και οι έχοντες προβλήματα σε αυτό το πεδίο θα εργαστούν άοκνα να υποστηρίξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτό το στόχο με επιτυχία. Ευχαριστώ. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρωτού δώσω τον λόγο στην εκπρόσωπο της ε, κυρίας της Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να πω ότι είσαστε στο σπίτι σας εσείς οι συντάκτες των αναφορών. Αυτό είναι το σπίτι σας και είμαι πεισμένος ότι η αναφορά που κάνατε πολύ καλά θα γίνει δεκτή από όλους τους ευρωβουλευτές. Είναι μια δίκαιη αναφορά αυτή πιστεύω και είναι μια αναγκαία αναφορά που πρέπει να ανταποκριθούμε στα αιτήματά της και είμαι πεισμένος ότι θα ανταποκριθούν οι ευρωβουλευτές σωστά στα αιτήματά σας. Είμαι πεισμένος γι' αυτό. Δίνω τον λόγο στη συνέχεια στην κυρία εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει τον λόγο παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συνεχίσω αγγλικά σας ευχαριστώ πολύ που προσκαλήσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενημερώσει για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ζήτημα αυτό, το οποίο συζητήθηκε και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Όπως υπόθηκε όντως, ο Επίτροπος Μπαρνιέ δεσμεύθηκε σαφώς απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να δοθεί εντολή στο Συμβούλιο να διαπραγματευτεί μια δεσμευτική διεθνή συνθήκη, συμφωνία, όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης. Προκειμένου όμως να εκπληρωθεί η δέσμευση αυτή, αυτό το οποίο άρχισε να κάνει ο Επίτροπος Μπαρνιά και οι υπηρεσίες του είναι να εγκριθεί καταρχά, καταρχάς μια σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για επίσημη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ζητήσει από το Συμβούλιο να δοθεί εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπραγματευτεί το διεθνές αυτό μέσο. Αν ζητάμε ουσιαστικά διαπραγματευτική εντολή, το κάνουμε γιατί θέλουμε μία νομικά δεσμευτική συμφωνία. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την εντολή αυτή, έχει εγκριθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων και θέλουμε να δοθεί λοιπόν η δυνατότητα από το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί το μέσο αυτό. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει συμβαλόμενο μέρος στο μέσο αυτό. Δεν μιλάμε μόνο για τα κράτη-μέλη, πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να αποτελέσει συμβαλόμενο μέρος. Να αποτελέσει συμβαλόμενο Έχει υποβληθεί λοιπόν στο Συμβούλιο το αίτημα αυτό. όπω είπε και η Κυπριακή Προεδρία έχει αρχίσει να συζητάτε το ζήτημα αυτό. Βλέπω ότι συμφωνούν και ορισμένα μέλη της ε, Επιτροπής σας. Όπως σας είπα, θα προτιμούσαμε να μπορούσαμε να λάβουμε πια άμεση με συγχωρείτε δράση, αλλά ουσιαστικά χρειαζόμαστε την υποστήριξη και την άδεια του Συμβουλίου προκειμένου να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε λοιπόν ακόμα μία επίσημη εντολή, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για μας. Χρειαζόμαστε στη διπλωματική διάσκεψη να έχουμε την επίσημη εντολή. Πρέπει αυτή να εγκριθεί λοιπόν το συντομότερο δυνατό, γιατί δεν μπορούμε να πάμε στη διπλωματική διάσκεψη χωρίς να έχουμε διαπραγματευτική εντολή στα χέρια μας. Στο ενδιάμεσο διάστημα όμως και στα πλαίσια της μόνιμης επιτροπής του WIPO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πολύ δραστήριο ρόλο, προσπαθώντας να καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί περαιτέρω εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που γίνανε πέρυσι και ανάμεσα στη συνεδρίαση αυτή και στην επόμενη που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα έχουν γίνει δύο άτυπες συνεδριάσεις όπου έχουν συμμετάσχει αρκετές χώρες συμπεριλαμβανομένων των μελών του WIPO που έχουν εκπροσωπηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία και προσπαθούμε στις συνεδριάσεις αυτές να ολοκληρώσουμε την εξέταση του κειμένου προκειμένου να διαθέσουμε το στομότερο δυνατό. Η τελευταία συνεδρίαση έγινε το Μάιο. Η, Επιτροπή, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γενέβη διοργάνωσε την συνεδρίαση αυτή. Γίνανε λοιπόν οι απαραίτητε συζητήσει προκειμένου να εξετάσουμε ορισμένε πτυχέ του κειμένου. Αυτά όσον αφορά την πρόοδο που έχουμε σημειώσει επί της ουσίας και με τις ίδιες προθέσεις θα πάμε στη Γενέβη την επόμενη εβδομάδα και ασκούμε πίεση αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο προκειμένου να έχουμε μία εντολή το στομότερο δυνατό, μία διαπραγματευτική εντολή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μαρτίν Πράτ. Να ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις. Η κυρία Βέρτμαν καταρχάς. Ε, ευχαριστώ, σας Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες, τους συντάκτες αναφοράς που είναι εδώ παρόντες. Ευχαριστώ και για την εικονική ανάγλυφη παρουσίαση για τους αριθμούς. 750.000 νέα βιβλία. Για να το δούμε αυτό και μόνο 30.750 για τους ε, έχοντες προβλήματα όρασης. Για να τα θέσουμε σε αναλογία αυτά, ίσως λέει, κάποια μέρα θα είναι στη διάθεση των ε, έχοντων προβλήματα όρασης. Διαρωτώ με πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και παιδεία, τι γίνεται με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρώπη και παγκόσμια να εκπαιδεύονται και να καλύπτουν τι ανάγκε του. Για τη συνάντηση στη Γενέβη την επόμενη εβδομάδα θέλω να θέσω το ερώτημα στο Συμβούλιο. Έθεσα ερώτημα στο Συμβούλιο σε σχέση με την εντολή. Θα ήθελα να μου πείτε παρακαλώ ποιες χώρες ακριβώς ε, έχουν προβλήματα σε σχέση με αυτή τη συνθήκη και τι μπορούμε εμείς πραγματικά ως Ευρωβουλευτές να κάνουμε ώστε επιτέλους πραγματικά να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Να υπάρξει δικαιοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με μας από ό,τι φαίνεται για τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόσα Βάγνερ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Τα άτομα τα οποία έχουν ε, προβλήματα όρισης ε, και η δυνατότητά τους να έχουν ε, ε, βιβλία είναι τμήμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης και επικύρωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, φέτος στην Ολομέλεια εγκρίθηκε ψήφισμα το οποίο απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό ε, τυφλών και άτομα με προβλήματα αναπηρίας και άλλες ε, δυσκολίες ανάγνωσης όπως είναι τα προβλήματα των ατόμων με δυσλεξία. Ε, ο επίτροπο Μπανιέ θα πρέπει να αποστείλει σαφέ μήνυμα για να διαπραγματευτούμε αυτή τη συνθήκη με σαφεί, αποτελεσματικού και χρήσιμου όρου. Σήμερα, αρκετού μήνου μετά και μετά ε, εν ώψη και της ε, διάσκεψης που θα γίνει στη Γενέβη την επόμενη εβδομάδα, δεν γνωρίζουμε ούτε την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε του Συμβουλίου. Θα υποστηρίξει μια δεσμευτική σύμβαση το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μόνο μια μορφή νομικού μέσου. Ε, η Ένωση για την ε, Πνευματική Ιδιοκτησία θα ζητήσει να υπάρξει μια διάσκεψη για να εγκριθεί συγκεκριμένη συνθήκη. Θα, ποιες είναι οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ε, διεθνή αυτή σύμβαση και οι θέσεις αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των τυφλών ατόμων να έχουμε ένα απλό μίγριο βραχικό κείμενο και αρκετά ασφαλές. Ζητάμε λοιπόν από την Κυπριακή Προεδρία που έχει την Προεδρία αυτή τη στιγμή του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δράσουν για ένα δέμα πολύ μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σόσα Βάγνερ, η κυρία Άουκεν στη συνέχεια. Yeah, ε, ε. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συναδελφοί μου. Και πρέπει να τονίσω επίσης ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια κράτη-μέλη μπλοκάρουν αυτή την πρωτοβουλία. Είμαι σε επαφή με την Δανέζικη κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προεδρίας τους κυρίως και αρχικά μας είχε δοθεί μια πολύ αρνητική εντύπωση ότι η γραφειοκρατία ήταν τέτοια σε επίπεδο Υπουργείου και δεν γνώριζαν ούτε καν ότι έπρεπε κάτι να κάνουν Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες εθελοντικές συμφωνίες κτλ. Και ουσιαστικά μας είπαν θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε κάτι τις συμφωνίες και να δούμε επίσης και τι συμβαίνει με την άκτα κτλ. Βέβαια, πρέπει να δούμε ότι δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια κατηγορία τα πάντα και έλαβα μια επιστολή από τη Δανέζικη κυβέρνηση πάλι πριν από μερικές εβδομάδες κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας και τότε έγινε μια αναφορά για μια δεσμευτική συμφωνία. Νομίζω λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο τις κυβερνήσεις και να τους πούμε ξεκάθαρα ότι ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ζούμε στον πεπαλαιωμένο κόσμο στον οποίο ζουν αυτοί, ότι έχουμε πλέον μια νέα πραγματικότητα στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε, ότι πρέπει να είμαστε σαφείς απέναντι στους πολίτες μας. Δεν μπορούμε να τους λέμε ότι δεν νοιαζόμαστε αυτή τη στιγμή για σας και ότι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η γραφειοκρατία κτλ. Δεν μπορούμε να λέμε στους πολίτες κατάφορα ότι δεν νοιαζόμαστε για εσά. Και αν υπάρχουν κάποιε κυβερνήσει που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κατανομαστούν. Σα eh, Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν θέλω καθόλου να επισέλθω στα θέματα ουσίας διότι είναι τόσο αυτονόητο αυτό το αίτημα και το ζήτημα. Η πρόσβαση στη λογοτεχνία και σε αυτά τα βιβλία πρέπει να διασφαλίζεται. Πρέπει υποχρεωτικά να διασφαλίζεται. Αυτό σήμερα υπό τα νέα δεδομένα των τεχνολογικών εξελίξεων είναι πολύ πιο εύκολο να διασφαλιστεί και επιτέλους να υπάρξουν ευκαιρίες για αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι σαφή. Τώρα το ότι τροχοπεδούνται αυτά τα πράγματα ότι δημιουργούνται προβλήματα από ανθρώπους που λένε ότι θα στείλουμε αυτές τις ενώσεις των τυφλών να διαπραγματευτούν για κάθε ξεχωριστό βιβλίο. Ε, αυτό είναι κινησμός, είναι αμοραλισμός. Για μένα αυτός είναι ένας κινησμός, ένας αμοραλισμός που δεν μπορώ να δεχθώ και να παρακολουθήσω. Είναι απαράδεκτος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια δεσμευτική συνθήκη, binding treaty. Δεν γίνεται καθόλου να έχουμε εθελοντικές, εθελούσιες συμφωνίες εθελοντικού χαρακτήρα. Δεν είναι το σωστό μέσο αυτό και δεν είναι διασυνοριακή δυνατότητα αυτή για την επίλυση του προβλήματος με κανένα τρόπο. Γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζω και να μου πείτε χαίρομαι επιτέλους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί αυτή την πορεία τώρα πια διότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να πιστεί, να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα έπρεπε να στέλνουν για διαπραγματεύσεις αιώνια ανθρώπους και να ζητούν να υπάρχουν αιώνια διαπραγματεύσεις. Χρειαζόμαστε ένα δεσμευτικό χρονοπλαίσιο. Πότε τι θα γίνει. Και επιτέλους χρειαζόμαστε και την, το να σταματήσει με τις διαπραγματεύσεις εν κρυπτό και παραβίστο το Συμβούλιο και να προστατεύει τα μέλη εκείνα του Συμβουλίου που προασπίζουν κάποια κεκτημένα του παρελθόντος και αν είναι δυνατόν με οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε γύρο διαπραγμάτευση δεν θέλουν να υπάρχει η δεσμευτική εντολή. Ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε ακριβώς ακολουθώντας τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου, πότε η επιθυμία προς το Συμβούλιο θα μπορέσει να προ... Ε, υποβλήθηκε για να διαμορφωθεί αυτή η εντολή. Και δεύτερο, προς το Συμβούλιο. Πότε συζήτησε αυτό το θέμα το Συμβούλιο και αν το συζήτησε με ποιο αποτέλεσμα, με, με ποια έκβαση. Να πείτε τα ονόματα, να κατονομάσετε τα κράτη εκείνα τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Πείτε το ανοιχτά και ειλικρινά. Ποιοι είναι που δημιουργούν προβλήματα. Έχω υποψίες εγώ για το ποια είναι αυτά τα κράτη. Αλλά θέλω να το πείτε εσεί καθαρά και ξεκάθαρα. Διότι αυτέ οι χώρε πρέπει να αποκαλυφθούν αυτές που λένε ότι τους είναι αδιάφορο αν υπάρχουν ε, προβλήματα για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης και τους είναι αδιάφορο και θέλουν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και για άλλα 50 χρόνια χωρίς θετική έκβαση, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Να μας πείτε ποια είναι αυτά τα κράτη επιτέλους. Και αν είναι αποφασισμένο το Συμβούλιο να διαπραγματεύεται και κλεισμένων των θυρών εγκρυπτό και παραβίστο, θα ξέρουμε ότι το Συμβούλιο είναι ανάξιο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Έγκστρομ τώρα. Ανώ, οκ. Okay. Antes de dar la palabra a los peticionarios... Ah, Ο κύριος Μποστινάρο πριν δώσει το λόγο στους αναφέροντες. And, uh, yeah, now it's, it's functioning. Ναι, λειτουργεί τώρα το μικρόφωνο. Ζήτησα το λόγο για να πω κι εγώ ποια είναι η άποψή μου για το ουσιαστικά να πω και την άποψή μου σε σχέση με τις πολύ σοβαρές παρεμβάσεις που κάνανε οι συνάδελφοι. Λάβαμε πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση και κάνει ουσιαστικά γρήγορα, επιτελεί γρήγορα το έργο της. Το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω προς την Κυπριακή Προεδρία καταρχάς και ξέρω ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν μπορεί να απορρίψει την όλη ιδέα ότι θα πρέπει να δοθεί μία μάχη για το ζήτημα αυτό. Δεν κάνουμε εδώ πέρα διαπραγματεύσει στα πλαίσια του Διεθνού ε, Νομισματικού Ταμείου. Δεν συζητάμε καν για το πακέτο συνοχή. Τα πράγματα είναι πολύ λιγότερο δραματικά από άλλα ε, δύσκολα ζητήματα. Θεωρώ ότι εδώ πέρα μπορούμε πολύ εύκολα να σημειώσουμε επιτυχία. Και Πιστεύω ότι η πρόεδρός μας, η κυρία Ματσόνη, θα πρέπει να αποστείλει μια επιστολή, γιατί ξέρουμε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι παρόν κάθε φορά στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισήμως να υποβάλει στο Συμβούλιο το αίτημα αυτό με τρόπο απολύτως ρητό ζητώντας από το Συμβούλιο να σταματήσει πλέον να ασχολείται κατά αυτό τον τρόπο με το πρόβλημα αυτό που έχει να κάνει ουσιαστικά με την τραγωδία που ζουν 500 εκατομμύρια άνθρωποι, που ουσιαστικά βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση εξαιτία των πνευματικών δικαιωμάτων να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια πνευματικά έργα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να ζητήσουμε από την Κυπριακή Προεδρία να δείξει σωστή καλή θέληση και βούληση να ασκήσει πίεση στα μέλη του Συμβουλίου και θα πρέπει επισήμω ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποβάλει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ το Συμβούλιο, προκειμένου το ζήτημα αυτό να αποτελέσει ζήτημα κατεπήγοντο, ζήτημα προτεραιότητο. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος κατά κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να βρεθεί στην πρώτη θέση για την προώθηση ενός ζητήματος που το παραλαμβάνω πιστεύω ότι μπορεί να επιληθεί εύκολα. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στους αναφέροντες, ε, διατυπώθηκαν πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Συμβούλιο για την ανάγκη να υπάρχει αυτή η δεσμευτική ε, συνθήκη. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου πρώτα. <clears throat> I believe, uh, before uh, giving us the floor... Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ετέθη ένα πολύ βασικό ερώτημα όσον αφορά την ε, εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως ήταν καλύτερο να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να απαντήσουμε εμείς στις ερωτήσεις. Um, to be very clear as to... Θα είμαι σαφής πώς εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Φεβρουάριο δεσμεύτηκε ο Επίτροπος Μπαρνιέ, συναντηθήκαμε μαζί του, ζήτησε από τις υπηρεσίες μας να συντάξουν την εντολή διαπραγμάτευσης. Αυτό έγινε σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία και σε διοργανική διαβούλευση και ουσιαστικά οι παρατηρήσεις που φτάσαν κατά τη διάρκεια τη διοργανικής διαβούλευση είχαν να κάνουν μόνο με τη βελτίωση του κειμένου, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 8η Ιουνίου, όταν ήταν έτοιμε και όλε οι, μετα... μεταφράσεις. Προχωρήσαμε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα, εφόσον πρόκειτο για απόφαση εντολής. Απεστάλλει λοιπόν το κείμενο αυτό στο Συμβούλιο και επιμένω ότι χρειαζόμαστε για τη διπλωματική διάσκεψη να έχουμε την εντολή αυτή. Γιατί χωρίς αυτή την εντολή δεν θα καταφέρουμε να διαπραγματευτούμε στην Γενέβη την επόμενη εβδομάδα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται αυτή τη στιγμή την υποστήριξη του Συμβουλίου σε αυτή τη φάση. Δεν χρειάζεται επίσημα τη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου προκειμένου να καταφέρει να διαπραγματευτεί στην Γενέβη την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ουσιαστικά ίσχυε και για τη συνεδρίαση η οποία έγινε και τον Νοέμβριο και σε όλες τις ενδιάμεσες διασκέψεις. Χρειαζόμαστε όμως πλέον να έχουμε αργά ή γρήγορα αυτή την έγκριση από το Συμβούλιο για την εντολή. Το λόγο έχει το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα πολύ βασικό αίτημα αυτή τη στιγμή να κατονομαστούν ουσιαστικά κάποια κράτη-μέλη. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το Συμβούλιο είναι συνομοθέτης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουσιαστικά βασιζόμαστε στη δική σας τη συνεργασία και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κατονομάσουμε αυτή τη στιγμή κράτη-μέλη. Μπορώ να σε εξηγήσω ότι έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά δεν μπορώ να αφαιρθώ τόσο πολύ στην υφιστάμενη κατάσταση. Στο παρελθόν, όπως το γνωρίζετε, υπήρχαν πολλά κράτη-μέλη τα οποία είχαν ενδιασμούς για να υποστηρίξουν ένα δεσμευτικό μέσο. Προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο δεσμευτικού νομοθετικού οργάνου, καταλαβαίνετε ότι απαιτείται πολύς χρόνος. Επομένως, είτε μας αρέσει ή όχι, ξέρω ότι εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να αναλώνω πάρα πολύ χρόνο για σημαντικά ζητήματα, Συμφωνώ πάντως με τη δική σας την στάση και καταλαβαίνω απόλυτα τις ανησυχίες σας και το ότι θέλετε να γνωρίζετε ποιος μπλοκάρει τι. Κανείς δεν μπλοκάρει όμως τίποτα. Αυτό το οποίο συνέβη, αυτή τη στιγμή είχαμε την εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Ιουνίου, η Προεδρία μας ε, ε ουσιαστικά ρυθμεί μόνο 11 μέρες αυτή τη στιγμή. Στις 4 ε, ε, Ιουνίου και στις 5 Ιουνίου ήμασταν στην Επιτροπή ε, νομικών θεμάτων και είπαμε ξεκάθαρο ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Και στις 5 Ιουνίου συγκεκριμένα συζητήσαμε το έγγραφο αυτό, το θέσαμε επιτάπητος στην ε, ομάδα εργασίας ε, του Συμβουλίου, στην αρμόδια ομάδα εργασίας και έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Και πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη, ουσιαστικά η πλειοψηφία των κρατών μελών, είχαν θέσαν επιφύλαξη, προτίμησαν να, επιστρέψουν στις πρωτεύουσές τους και να ζητήσουν μία ξεκάθαρη εντολή από τις υπηρεσίες τους προκειμένου να γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν στην επόμενη ομάδα εργασίας. Το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί το Σεπτέμβριο, στις 13 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ε, αρμόδιας ομάδας εργασίας του Συμβουλίου. Τώρα όσον αφορά το ποιος απορρίπτει την όλη πρόταση και όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία. Θα κάνουμε κάθε το δυνατό για να προωθήσουμε το ζήτημα. Ξέρετε ότι και για μας αποτελεί προτεραιότητα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της εξάμενης προεδρίας μας. Σας διαβεβαιώ και το λέω αυτό ξεκάθαρα εδώ, ότι θα κάνω κάθε τι το δυνατό ως προεδρεύουσα της αρμόδιας ομάδας εργασίας συμβολίου προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα με παρούσα και στις συζητήσεις που θα γίνουν στο CCR και αυτό αποτελεί επίση απόδειξη ότι λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μα το ζήτημα. Σε κάθε πάντως περίπτωση υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να έρθουμε σε επαφή με τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν εκφράσει ενδιασμούς και σκεπτικισμό. Όπως σας είπα όμως, ε, τα κράτη-μέλη, κανένα κράτος μέλος δεν εξέφρασε σκεπτικισμό για να συζητήσουμε το, μάλλον για τη δυνατότητα να υπάρξει δεσμευτικό όργανο στις 5 Ιουνίου. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά κράτη-μέλη τα οποία λέγανε ότι δεν θέλουν δεσμευτικό όργανο. Αυτή τη φορά δεν το απορρίψανε. Είχαν απλώς μια επιφύλαξη μελέτης προκειμένου να συζητήσουν περισσότερο με τις πρωτεύουσέ τους και να καταφέρουν να δώσουν την πραγματευτική εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί όπως βλέπετε. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεσμεύομαι θα κάνω κάθε το δυνατό για να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Χόκεν είχε ζητήσει τον λόγο. Παρακαλώ πολύ σύντομη παρακαλώ για να πάρουν τον λόγο οι συντάκτες της αναφοράς. Θα είμαι πολύ σύντομη Ξέρω ότι δεν είναι θέμα συναπόφαση εδώ. Όταν είπατε όμως ε, συναπόφαση, συνομοθεσία και είπατε να μην κατονομάσετε τα κράτη αυτά, θέλω να σα πω ότι έχουμε διαφάνεια στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν συνεργάζεστε μαζί μα και εσεί ε, πρέπει να διασφαλίζετε την διαφάνεια. Ξέρω ότι κάποιοι δεν ικανοποιούνται ιδιαίτερα με αυτό από πλευρά του Συμβουλίου, αλλά αυτό πρέπει να συμβαίνει. Δημοκρατία και διαφάνεια απορρέει και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πείτε λοιπόν παρακαλώ στα μέλη του Εξαιρετικού Συμβουλίου ότι θα θέλαμε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και ξέρουμε όλοι από όλα τα κράτη-μέλη μας ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους τα μέλη του Συμβουλίου και υπάρχουν δυσκολίες και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν μέσα άσκησης πίεσης να προχωρήσουν. Ευχαριστώ που το σχολιάσατε αυτό. Uh, sorry, ε, ε- Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Εγώ δίνω τον λόγο αν συμφωνείτε. Έχετε τον λόγο τώρα <laughs> να συνεχίσετε. Μάλιστα είναι η πρώτη μου φορά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο γι' αυτό. Είναι τα πρώτα μου βιώματα αυτά. Είμαι αρχάρια, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, δεν εννοούσα ότι δεν είσαστε συνομοθέτες Τούτου καθέντος, φυσικά επειδή υπάρχει η συνθήκη τη Λισαβόνα και επειδή κατανοώ απόλυτα όλα αυτά τα θέματα, νομοθετούμε για του πολίτε και εσεί είσαστε υπεύθυνοι αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών και είναι πολύ σημαντικό για εσά να γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτά τα θέματα στα οποία εμπλέκεστε και γι' αυτό το είπα αυτό το οποίο είπα και γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ σήμερα για να παρακολουθήσω είναι ένα διεθνέ μέσο αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά δεν έχει δικαιώματα να ψηφίσει επ' αυτού. Όμως είμαστε εδώ να επεξηγήσουμε, να σας συναντήσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αυτές τις επαφές ε, και πιο, σε πιο άτυπο πλαίσιο ώστε να προαχθεί το θέμα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουν τον λόγο οι συντάκτες της αναφοράς παρακαλώ. Um... Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όμως οι συζητήσεις που ακούσαμε, οι παρεμβάσεις και επεξηγήσει του Συμβουλίου και τη Επίτροπή, που ήταν βέβαια πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά οδηγούν σε τρεις παρατηρήσεις που θα ήθελα να ζητήσω αποσαφηνήσεις επ' αυτών. Είναι πολύ πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο μόλις, που οι διαπραγματευτέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότειναν ένα μέσο που να εξυπηρετεί αυτό το στόχο και πρότειναν να μην είναι δεσμευτικού χαρακτήρα, να είναι ήπιο νομοθετικό έργο. Αυτό όμως είναι στο ιστορικό πλαίσιο, στο παρελθόν πια. Αυτά όμως μας ανησυχούν κάπως και θέλουμε τώρα πια να έχουμε μια σαφή ένδειξη από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα είναι δεσμευτικού χαρακτήρα αυτό το μέσο Ξέρουμε ότι ε, καταβάλει προσπάθειες ο Επίτροπος και το Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες και αυτό που αναφέρθηκε υποστηρίζει ακριβώς ε, σε σχέση με τον κύριο Μπαρνιέ που θέλει να υπάρξει μια δεσμευτικού χαρακτήρα συνθήκη. Μετά ακούμε τον όρο νομικό μέσο και όχι δεσμευτική συνθήκη. Είπατε ότι αναφέρεστε στο ίδιο πράγμα και θα είναι το ίδιο, όμως εμείς θέλουμε να είναι μια δεσμευτική συνθήκη, δεδομένη της προϊστορίας όμως και μια και θέλουμε να υπάρχει μια δεσμευτική συνθήκη ούτως ή άλλως θα μας διασφάλιζε τα συμφέροντά μας αν αναφερόταν αυτό ως δεσμευτική συνθήκη και όχι ως κάτι άλλο. Λοιπόν, αναζήτησε κάποια εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια δεσμευτικού χαρακτήρα συνθήκη. Θα ήταν χρήσιμο αν θα μπορούσατε να πείτε δεσμευτική συνθήκη και τίποτα άλλο. Και για την κυρία Μαρτίν Πράτα διευκόλυνε τα πράγματα. Δεν θα ζητούσαμε διαρκώς να μας διασφαλίζει ότι θα γίνονται διαπραγματεύσεις για μια δεσμευτικού χαρακτήρα συνθήκη, αν αυτό διασφαλιστεί εξάπαντος. Και το θέμα για την διπλωματική διάσκεψη. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο όταν καταλήγει κανείς σε μια διπλωματική διάσκεψη, τότε χρειάζεται αυτό το μέσο της ε, ε, δεσμευτικού χαρακτήρα συνθήκης Στι διαπραγματεύσει μπορούν να διαπραγματεύονται διαφορετικά. Το κατανοώ αυτό. Αν όλοι όμως ε, πιέσουν και ζητήσουν να διεξαχθεί μια τέτοια διπλωματική διάσκεψη το 2013 και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει ακόμα ένα μέσο για μια δεσμευτικού χαρακτήρα συνθήκη θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέση να δεχθεί από κοινού με τα άλλα κράτη-μέλη και να πει ότι μάλιστα ναι, θα επιτρέψουμε να διεξαχθεί μια τέτοια διπλωματική συνθήκη για να δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη. Παρότι η Επιτροπή δεν θα έχει τις επόμενες δύο εβδομάδες αυτή την εντολή. Και θα ήθελα εν τέλει, τελευταίο σημείο, μια διευκρίνηση για τον Επίτροπο Μπαρνιέ που είπε ότι θα έρθει σε επαφή και θα διαπραγματευτεί με κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος που ακούσαμε να παρουσιάζεται, είναι κάτι που θα το κάνει μετά από αυτή τη συνάντηση ή όχι. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω τώρα ότι θα επιτρέψετε να υποβάλω μια πρόταση που είναι αρκετά απλή οι συντάκτες αναφοράς κατάφεραν πιστεύω να διαπιστώσουν ότι υπάρχει ομοφωνία στα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής για να ζητήσουμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο το δυνατόν πιο γοργά να καταλήξουμε σε μια ε, συνθήκη δεσμευτικού χαρακτήρα. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου και νομίζω ότι ήταν θετική αυτή η πληροφόρηση που μας έδωσαν Συγκεκριμένα η Κυπριακή Προεδρία που έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διασφάλισε ότι είναι ένα θέμα ύψης της προτεραιότητας και έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε και να ολοκληρώσουμε στη γραμμή της πρότασης που έκανε ο κύριος Μποστινάρ ότι η Προεδρία αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με επιστολή θα στραφεί <clears throat> στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Κυπριακή Προεδρία και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβιβάζοντας και λέγοντας ότι ομόφωνα η Επιτροπή Αναφορών ομόφωνα ζητεί απαιτεί, διεκδικεί να μην υπάρξει καθυστέρηση. Να μην υπάρξει καθυστέρηση ώστε να δημιουργηθεί άμεσα μια δεσμευτικού χαρακτήρα συνθήκη για να επιληθούν αυτά τα οποία εμεί θεωρούμε <clears throat> ε, τα θέματα ε, ισότητας ε, επί των αρχών ισότητας δικαιωμάτων των πολιτών να διασφαλίζεται ότι αυτές οι ενώσεις και σύλλογοι και εκείνοι των μειονεκτούντων ατόμων που έχουν τη μειονεξία της δυσλεξίας και οι άλλοι να έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην δυνατότητα ανάγνωσης όπως όλοι οι πολίτες ανάγνωσης βιβλίων. Και είναι ομόφωνη η θέση των μελών της Επιτροπής μας και με επιστολή θα μπορέσουμε να διαβιβάσουμε αυτές τις θέσεις στα τρία θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είσαστε υπέρ αυτής της πρότασης. Παρακαλώ. Ναι, εσείς κύριε συντάκτη αναφοράς έχετε τον λόγο κύριε εκπρόσωπε των αναφερών. Thank Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η υποστήριξη της οποίας τύχαμε σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή από τους Ευρωβουλευτές, από το Ευρωκοινοβούλιο. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις απαντήσεις στις τρεις ερωτήσεις που διατυπώσαμε, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν ήδη την επόμενη εβδομάδα στη Γενέβη για αυτά τα θέματα. Και θέλουμε να δούμε μια και γραπτέ ανταλλαγές και πληροφόρηση γραπτή διεπιστολή δεν θα μπορέσει να καλύψει αυτά τα μικρά χρονικά διαστήματα. Να μας δοθούν απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία διατυπώσαμε. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Όσον αφορά την ε, γλώσσα, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όταν ζητάμε μία εντολή, ακολουθούμε ακριβώς το θεσμικό σύστημα το οποίο προβλέπεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μία εντολή προκειμένου να διαπραγματευθεί μία τέτοια συνθήκη. Όταν όμως χρειαζόμαστε μία απόφαση για διεθνή συμφωνία, και όταν γίνεται σύσταση προς το Συμβούλιο για να υπάρχει μια διαπραγματευτική εντολή, τότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και ως προς αυτό θα έλεγα προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τι θα γίνει τώρα στο SSER, πολύ καλό το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για διπλωματική διάσκεψη βρίσκεται στα χέρια της Γενικής Συνέλευσης της Γενέβης. Αν όλα πάνε λοιπόν κατευχήν και αν όντως δούμε ότι θα επιτευχθεί η απαραίτητη πρόοδος, τότε θα ληφθεί μία απόφαση από τη Γενική Συνέλευση της Γενέβης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως, εφόσον προκύψει αυτή η δυνατότητα, θα κάνει κάθε το δυνατό προκειμένου να δοθούν αυτές οι απαραίτητες συστάσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να επισημοποιηθούν μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή όμως να πω παραπάνω πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επιβάλλει τίποτα στα κράτη-μέλη, ούτε μπορεί να μιλήσει εξ ονόματος των κρατών μελών. Χρειάζεται την υποστήριξη των κρατών μελών. Όσον αφορά τη δέσμευση του Επιτρόπου Μπαρνιέ, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και αυτό που έχει κατά νου άλλωστε ο κύριος Μπαρνιέ και το έχει πει και άλλωστε πολλές φορές, είναι ότι δεν θα είναι καλή ιδέα και δεν θα είναι αποτελεσματικό να πρέπει να πάει σε κάθε ένα από τα, κράτος μέλο, σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη ξεχωριστά. Θα χρειαστεί να αναλώσει πάρα πολύ χρόνο και προφανώς έχει και άλλες υποχρεώσεις. Είμαι πάντως πεπισμένη ότι ε, θα πάρει το λόγο και θα μιλήσει δυναμικά αν τυχόν υπάρξει αντίδραση ή αντίσταση από συγκεκριμένα κράτη-μέλη όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε κυρία Μαρτίν Πράτ. Επαναλαμβάνω λοιπόν την πρόταση που σας έκανα, που νομίζω ότι είναι και η αίσθηση της πλειοψηφίας, αν όχι του συνόλου των μελών της Επιτροπής, να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους αναφέροντες, διότι μπορέσαμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτή την ομάδα ανθρώπων που είναι τόσο σημαντική και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Νομίζω ότι έχουμε ομόφωνη υποστήριξη από όλου και θα προσπαθήσουμε να σα βοηθήσουμε να βρείτε... Ε, υποστηρικτέ, ένθερμου και εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φυσικά και του Συμβουλίου. Και ολοκληρώνεται το ζήτημα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.